Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne euh, journée. Nous allons commencer... Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Καταρχάς, κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχά, σε σχέση με την ίδια διάταξη, το σημείο 8 θα συζητηθεί μετά το σημείο 3, το σημείο 9 μετά το σημείο 7 και το 5 μετά το 9. Le point. Τα 18 και 19. Μετά το 22. Να τα επαναλάβω, μήπως. Λοιπόν, το 8 μετά το 3. Το 9 μετά το 7. Το 5 μετά το 9 και τα σημεία 18 και 19 μετά το 22. Υπάρχει αντίρρηση, απορία. Αν όχι, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι εγκρίνεται λοιπόν η για διάταξη. Και έρχομαι στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Επειδή έχω ένα πρόβλημα στο αριστερό μάτι και δεν μπορώ να διαβάσω ε, το κείμενο που είναι πυκνογραμμένο. Θα παρακαλέσω την γραμματεία. Αλλά σε 15 ημέρες μετά την χειρουργική επέμβαση θα είμαι καλά. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας και παρακαλώ τη γραμματεία να διαβάσει λοιπόν, σχέδιο εκτελεστική δράση για τον κανονισμό 2007-2001 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου υπευλήθη τέλη Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για μια εκτελεστική πράξη με στόχο την επικαιροποίηση υφιστάμενης εκτελεστικής πράξης για να ληφθεί υπόψη η κωδικοποίηση του βασικού κανονισμού του περσινού έτους. Ε, δεδομένης της αίτησης της Κομισιόν να αντιμετωπιστεί κατεπηγόντως το θέμα, ο μόνιμος εισηγητής για την επιτροπολογία και την εκχώρηση νομοθετικών εξουσιών κ. Γιάννης Ρόντε προτείνει κατ' εξαίρεση να γίνει γραπτός η εξέταση από την Επιτροπή μας προκειμένου να εγκριθεί και να τεθεί σε ισχύ η επικαιροποιημένη εκτελεστική πράξη το συντομότερο δυνατό. Δεν ε, κάποιο δεν λήφθη κάποιο σχόλιο από τους βουλευτές. Επομένως, δεν θα γύρει ενστάσεις στο Κοινοβούλιο δυνάμει του δεδομένου εξέτασης που προβλέπει το άρθρο 11 του κανονισμού που αφορά τις, αφορά δράσει δράσεις, σχέση με τη συγκεκριμένη πάντα. Εκτελεστική πράξη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λέω πρόεδρος, αν δεν έχω λάβει αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 22ης Νοεμβρίου 2017 και της 15ης Ιανουαρίου 2018 θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της κυρίας Μπερζεγόν. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Ε, ε mes chers Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία μικρή παρένθεση σε σχέση με τις γονικές άδειες, ε, γιατί μας έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις. Ε, στις 16 Φεβρουαρίου ε, η Microsoft είπε ότι θα δίνει τις ίδιες γονικές άδειες σε σε όλο τον κόσμο, 20 ε, εβδομάδες για τις γυναίκες και 6 εβδομάδες για τους άντρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος κοινωνική, ε, γιατί μπορεί αυτό να έχει αντίκτυπο και στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι οποίες βρίσκονται πολύ κάτω από αυτά τα όρια αγωνικής άδεια. Θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και αναφέρομαι κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτή την οικονομική προσπάθεια. Όμως είναι ένα μήνυμα πολύ ισχυρό, ε, το οποίο πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο κείμενο λοιπόν που εξετάζουμε σήμερα, η οδηγία που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να αντιμετωπίσει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να υποστηρίξει την ε, ε, πρόοδο της καριέρας τους στι στις ίδιες συνθήκες εξισορρόπησης οικογενειακού και ιδιωτικού βίου. Ε, συμφωνούμε όλοι με αυτό το στόχο βεβαίως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις διάφορες τροπολογίες που καταθέσατε ε, που συμμετέχουν σε αυτή τη λογική και δίνουν, ε, βελτιώνουν την, ε, την ε, σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα του ε, κειμένου. 63,4% ε, από 20 έως 64 ε, ε, ετών είναι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Η, η διαφορά ακόμη στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι έντονη, ειδικότερα για τους γονείς και για όλους όσους έχουν άλλου είδους οικογενειακές υποχρεώσεις. Η αιτία είναι οι ανεπαρκείς πολιτικές εξισορρόπησης επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Όπως γνωρίζετε, οι εθνικές νομοθεσίες σχετικά με το θέμα αυτό ποικίλουν και προβλέπουν λίγες διατάξεις ε, για να αναλάβουν ισότιμα τις ε, οικογενειακές ευθύνες οι άντρες δίπλα στις γυναίκες. Ε, πιστεύω ότι η πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθεί να καλύψει τα κενά αυτά. Σε γενικέ γραμμέ, συμφωνώ με την πρόταση, τη θεωρώ ότι αποτελεί μια κοινωνική πρόοδο, όμως διαβάζοντας ε, τις τροπολογίες τους βλέπω επίσης ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις ή συμπληρώσεις που είναι απαραίτητες όσον αφορά την, την ηλικία των παιδιών, τις προθεσμίες των γενικών αδειών ε, ή τον χαρακτήρα υποχρεωτικό ή μη των ε, αδειών πατρότητας. Τέσσερα λοιπόν σημαντικά ζητήματα, γονική άδεια, ε, άδεια πατρότητας, ε, ευέλικτες μορφές εργασίας ε, και αμοιβή. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφερθώ ξεχωριστά σε αυτά τα στοιχεία όσον αφορά την άδεια πατρότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει την εισαγωγή ενός δικαιώματος 10 αμοιβόμενων ημερών εργασίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πιο πέρα και να το καταστήσουμε αυτό υποχρεωτικό, αμοιβόμενο, ώστε να δείξουμε έντονα ε, να προωθήσουμε σε έντονο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και έτσι θα μοιάζονται το άχθος ε, ε, του να είναι κανείς γονέας εξίσου οι άντρες και οι γυναίκες. Και θα ενθαρρύνουμε τη σχέση πατέρα και παιδιού. 11 ημέρες είναι σε μερικές χώρες οι, ε, οι άδειε αυτές, όμως είναι διαφορετική κατάσταση σε άλλες χώρες. Μία μέρα στην ε, Γερμανία, ε, μία μέρα στην Ελλάδα, καμία στην Ιταλία. Διακόπτει ο πρόεδρος. Μήπως μπορώ να σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο αργά. Μα προσπαθώ, λέει η ομιλήτρια. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι ολυμπιακό άθλημα η διερμηνία. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η άνηση, με, η άνηση ε, αντιμετώπιση των γονεϊκών ευθυνών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών έχει ως αποτέλεσμα ότι οι γυναίκες ε, ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά με τους άνδρες γιατί δεν έχουν ε, καθόλου χρόνο άδειας, κάτι το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση και ως προς την εξισορρόπηση οικογενειακού και ιδιωτικού βίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια συμβιβαστική τροπολογία ω προ την άδεια πατρότητα ε, για να μπορείτε κι εσείς να μπορούν να ληφθούν υπόψη ευαισθησίε για το θέμα αυτό αυξάνοντα την διάρκεια τη άδεια πατρότητα ε, και καθιστώντα την αμοιβόμενη και υποχρεωτική. Στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ούτε και στι τροπολογίε, δεν υπάρχουν ε, σχετικά στοιχεία με τι πολλαπλέ υιοθεσίε και τι γεννήσει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι όλο και περισσότερε πολλαπλές γεννήσει υπάρχουν στις κοινωνίε μας. Νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το θέμα και να προβλέψουμε την αύξηση, ε, την επέκταση των γονεϊκών αδειών ε, λόγω του φαινομένου αυτού. Το προτείνω στην τροπολογία 10 και θα ακούσω και τις δικές σας απόψει όσον αφορά τώρα τη γονεϊκή άδεια. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να θεωρηθεί ε, το δίκαιο σε αυτή τη στιγμή, ώστε να είναι ευέλικτη άδεια τέσσερις μήνες μη ε, μεταβιβάσιμους και μη αμοιβόμενους. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη την ηλικία του παιδιού. Είναι κάτι που αναφέρεται σε όλες τις τροπολογίες σας. Ότι μπορεί δηλαδή κανεί να πάρει άδεια ε, γονική μέχρι τα 13 και όχι μέχρι τα 12, όπω λέει η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το αγγλοσαξονικό σύστημα που ε, όλοι το καταλαβαίνουν αναφέρεται σε teenagers, σε έφηβο, όχι 13 δηλαδή, 13 ετών, 14 ετών εγώ είμαι κάπως επιφυλακτική στη μείωση της ε, ηλικία, όπως προτείνει η κυρία Φεραγκούτη ο κύριος Άντερσον, γιατί νομίζω ότι δεν ε, θα επέτρεπε την ε, καλύτερη επιστροφή στην αγορά εργασίας των γονέων. Επίσης, το, το, η γονική άδεια καλό είναι να λαμβάνεται όταν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία. Ε, και μάλιστα εσείς προτείνετε 8 έτη, δεν την κατάλαβα αυτή την πρότασή σας. Κυρία Μερεγκό, το κύριος Μαρίνο και ε, ο κύριος Μπούντα ε, έχουν ε, καταθέσει τροπολογίε σε σχέση με το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η διάρκεια τη άδεια πρέπει να αυξηθεί για, τα, ε, παιδιά με, για τους γονείς παιδιών με αναπηρίε ή με σοβαρή ασθένεια. Το θέμα είναι, θα διπλασιάσουμε αυτήν την διάρκεια ή απλώ θα περάσει από 4-6 μήνε. Το ίδιο ισχύει και για τους μόνους γονείς, θα το συζητήσουμε. Ένα ακόμη ερώτημα για τον κύριο Μαρινό, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν προβλήματα ορολογία και μετάφραση των Ιταλικών στα Πορτογαλικά. Ε, αναφέρεστε στους ε, εργοδότες και στους άλλους εργαζομένους. Θα μπορούσαμε να πούμε και μισθωτούς. Εσείς χρησιμοποιείτε συστηματικά τον όρο εργαζόμενοι και δεν αναφέρεστε σε κανέναν άλλον όρο. Στα χαλικά είναι μια κατηγορία κοινωνική πολύ πιο περιοριστική από αυτή των εργαζομένων ε, που μπορούν επίσης να είναι μισθωτοί. Από ό,τι κατάλαβα, με τον όρο εργαζόμενοι λέτε και τους εργοδότες. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τη διάρκεια μεταξύ αυτών δύο κατηγοριών. Εργαζόμενοι, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αν χρησιμοποιούμε το ρόλ, τον όρο ε, εργαζόμενος στα γαλλικά. Όσον αφορά τώρα το δικαίωμα των γονέων για την, ε, για, την αμοιβή, ο πατέρα, συνήθως που παίρνει τον υψηλότερο μισθό μεταφέρει το δικαίωμα της άδεια στη γυναίκα γιατί αμείβεται λιγότερο ή καθόλου και αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια έχει μικρότερο εισόδημα. Πολύ λίγοι πατέρες παίρνουν την άδεια αυτή, 2,7%. Στη Γαλλία πάνω από 5% και το θέμα της, με, της μεταβιβασιμότητας και της αμοιβή ε, είναι το επίκεντρο του προβλήματος. Μπορεί αυτό να στοιχήσει πολύ στους εργοδότες και πρέπει να τους ε, προστατεύσουμε με ε, εγγυήσει ευελιξίας για να μπορέσει να υπάρξει συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Αυτή η οδηγία δεν πρέπει να αποτελεί ένα πρόβλημα και ένα εμπόδιο στις μικρές και πολύ μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. δεν πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον διοικητικοί περιορισμοί. Πρέπει να υπάρξει συνεπώ μια ισορροπία για να υπάρξει ένα, ένα ελάχιστο σύστημα αλληλεγγύη κοινωνικό. Είναι απαραίτητο για τι γυναίκε, δεν χρειάζεται να γίνουν φτωχότερε επειδή ε, κάνουν οικογένεια. Είναι, ε, ε, επίσης συμφωνώ ότι τουλάχιστον τρει μήνες δεν πρέπει να μεταφέρονται στον άλλο γονέα, γιατί είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Αν πρέπει να υποχρεώσουμε τους πατέρες να πάρουν αυτή τη γονική άδεια ε, για τις ευθύνες τους. Ε, ε, και συμφωνώ με τους, ε, με συναδέλφους που έκαναν σχετικές τροπολογίες που προτείνουν έναν μόνο μήνα και νομίζω ότι αυτό ε, δεν θα είναι αποτελεσματικό. Όσον αφορά τώρα την άδεια ασθενεία. πιστεύω ότι η αμοιβή πρέπει να είναι επαρκής και όχι απλώς συμβολική. Νομίζω ότι το να συνδέεται με, το, με τις ημέρε που δεν εργάζεται κανεί είναι το ελάχιστο. Επίση πρέπει να μπορεί ο εργοδότης να το αναβάλει το το χρονικό διάστημα της άδεια για ένα εύλογο χρονικό διάστημα αν θεωρεί ότι αυτό θα ε, δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στη συνέχιση της δραστηριότητας επιχείρησης. Καταλαβαίνω. Αλλά γιατί 20 μέρες. Γιατί έχετε διαλέξει τις 20 μέρες. Είναι 20 μέρες εργάσιμες ή 20 ε, μέρες... Ε, ε, συνεχείς διαδοχικές. Για τις πέντε ημέρες ε, ε, άδειας που προτείνεται, συμφωνούμε ότι πέντε, πέντε μέρες το χρόνο δεν είναι ε, επαρκής, όπως κύριε Κεσβαρά, Ροζιέρ, Κρυσόγονος ε, ε, και Μαστάλκα, ε, ζητούν να αυξηθεί αυτό το διάστημα και θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό. Επίσης πιστεύουμε όμως ότι αν αυξηθεί, αυξηθεί επικουρική άδεια, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα ε, για τον εργοδότη και την ε, λειτουργία της επιχείρησης. Ε, είμαι λοιπόν κάπως επιφυλακτική ως προς τις τροπολογίες Χρυσόγονου και Χάουταλα για το θέμα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διατηρήσουμε ε, την ιδέα της ανωτέρας βίας, ε, των ε, επιγουσών περιπτώσεων οικογενειακής, οικογενειακών έκτακτων καταστάσεων και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απουσίας από τη δουλειά για λόγους ανωτέρας βίας από τη στιγμή βέβαια που υποβάλλονται και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία η εισαγωγή της μεθόδου ευέλικτης εργασίας δίνουν τη δυνατότητα ε, στους γονείς μέχρι την ηλικία των 12 ετών να προσαρμόζουν τα ωράρια εργασίας τους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό στοιχείο αυτής της οδηγίας και θα δημιουργήσει καλύτερη ισορροπία οικογενειακού και ιδιωτικού βίου, ε, θα καταπολεμήσει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό να δοθεί δυνατότητα στον εργοδότη να ζητήσει περισσότερο στον ε, εργαζόμενο συγγνώμη, περισσότερες, περισσότερη ευελιξία στον εργοδότη ε, και υπάρχει ανάγκη γραπτής απάντησης ε, όταν αρνείται ο εργοδότης αυτήν την ευέλικτη εργασία. Νομίζω επίσης πρέπει να τους καθησυχάσουμε ότι θα ξαναβρούν τη θέση εργασίας τους όταν γυρίσουν από τη γονική άδεια πατρότητας ή μητρότητας, ισορροπία μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων και των εργοδοτών και υποστηρίζω τις τροπολογίες 134 και 146 του κυρίου Μπουντά, 144 ε, της Χάουταλα, 147 Ρέγνερ, 141 Μαρίνο, 158 ε, Κασπαρά και Ροζιέρ. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Χρυσόγονο, ε, αλλά ξέρω ότι έρχεται σήμερα το απόγευμα, και, ο κύριος Μαστά, και τον κύριο Μαστάλκα για την 149 όσον αφορά ε, την άρνηση ευέλικτης εργασίας και το εύλογο χρονικό διάστημα υποβολής των στοιχείων. Δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί περισσότερη σαφήνεια σε σχέση με την παράγραφο 2, την οποία αφορά ε, κυρία Ροζιέρ και Γκασμπαρά στην 151 τροπολογία σας για το άρθρο 13 παράγραφος 1 προσθέτεται ότι η δικαστική ε, απόδοση της άδεια ε, πρέπει να γίνεται ε, με μια ταχύτερη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούν να εγγυηθούν τέτοιου είδους διαδικασία. Η εμπειρία μου στα νομικά ζητήματα μου έχει δείξει ότι χρειάζονται ευέλικτοι κανόνες και νομοθεσίες, απλά πλαίσια και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να αποτελεί πάντοτε γνώμονα για τις δράσεις μας. Ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για το δικαίωμα των εργαζομένων 71, 117, 118 του κυρίου Χρυσόγονου ή για το δικαίωμα των ε, ασθενών 158 ε, της κυρίας Ρωσιέρ νομίζω ότι πηγαίνει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, υπερβολικά πολλές ε, γιατί το νομικό πλαίσιο εξελίσσεται βάσει αυτής της ε, οδηγίας ε, που σκοπό έχει να υπάρξει καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακού και ιδιωτικού βίου μεταξύ των γονέων και των φροντιστών και να τους δώσει συγκεκριμένα δικαιώματα όπως και συγκεκριμένα δικαιώματα στους ασθενείς. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι τελευταίο. Είμαι επιφυλακτική για την τροπολογία νέας, ε, για τη νέα νομική βάση για το κείμενο αυτό και μιλάω για την 28 του κυρίου Χρυσόγονου, 50 Γκασμπαρά και Ροζιέρ που αναφέρονται στα άρθρα 151 και 157 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το 153 άρθρο είναι η νομική βάση. Νομίζω ότι αυτό δεν συνεισφέρει στη σαφήνεια του κειμένου. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και άλλα σημεία ε, τα οποία ε, δεν θα τα θέσω γιατί έχω ήδη μιλήσει πάρα πολύ ώρα και θα μιλήσω ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά το προσωρινό χρονοδιάγραμμα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 29 Μαρτίου αυτό προβλέπουμε με τη γραμματεία. Θα μπορέσουμε να βρούμε, πιστεύω, συμφιβασμούς. Ε, θα το συζητήσουμε και με email μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και μου. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε βέβαια και να οργανώσουμε και επίσημες συναντήσεις με τους σκιώδους ε, εισηγητέ. Σας αφήνω λοιπόν το λόγο για να ε, με σχολιάσετε. Euh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το συγκριτικό πλαίσιο, ε, ιδιαίτερα περίπλοκο, σε σχέση με την εξισορρόπηση μεταξύ ιδιωτική και επαγγελματική ζωής. Θα αρχίσουμε με την κυρία Κάουφμαν. Ανοίγει η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να ζητήσω ε, συγγνώμη γιατί ο συνάδελφος ε, δεν είναι ε, εδώ, τον οποίο περίμενα και γι' αυτό δεν θα μπορέσω να απαντήσω όλες σας τις ερωτήσεις σας, αλλά θα σας παρουσιάσω ε, αυτό που υποβάλλει ο ίδιος, ο Ενρίκε Γκασπάρ. Ευχαριστώ πολύ για τη γνωμοδότηση της εισηγήτριας, γιατί καλύπτει πολυπληθείς προτεραιότητες ύψης της σημασίας για την ομάδα μας, ε, όπως η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η ισότητα ιδιωτική και επαγγελματικής ζωής, πολέμηση της περιθωριοποίησης και ιδιαίτερα των γυναικών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας. Θα πρέπει να ε, να προωθούμε την επανέμνωση της οικογένειας, δίνοντας κίνητρα για την συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών που εργάζονται. Όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες, θα πρέπει να τις λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περίπτωση, για αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας. Έχουμε 165 τροπολογίες. Θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, μίλησαν για αύξηση των αδειών, ιδιαίτερα για οικογένειες με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επεκταθεί η άδεια για τους φροντιστές τις 10 ημέρες το χρόνο. Σε σχέση με την παραβίαση των συνθήκων χορήγησης ε, άδεια, θα πρέπει να υπάρχουν αποτρεπτικές κυρώσεις έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ε, επιλογής ένδικων μέσων. Οι νέες ευρωπαϊκές κοινωνικές προκλήσεις θα πρέπει να πληρωθούν όσον αφορά την προστασία δικαιωμάτων και καταπολέμηση διακρίσεων καθώς και την πρόθεση των ε, συνθήκων εργασίας των εργαζομένων. Ως προς τις άδειες θα πρέπει να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή μεταξύ των θέσεων που έχουν υποβληθεί αλλά για να φτάσουμε σε μια πραγματική συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και για να φτάσουμε σε μια μακροχρόνια στρατηγική θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια συμφιλίωσης ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Θα πρέπει να τονίσω δύο ζητήματα που είναι ύψη τη σημασίας για μένα. Καταρχήν η επανακατανομή άδεια με νέες μορφές ε, που προτείνονται στην ε, τροπολογία 128 και την μη μεταβιβασιμότητα της ε, άδεια πατρότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από την ομάδα μου υπάρχει η θέληση να φτάσουμε σε ένα συμβασμό όλων των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χαουτάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι με εκπλήσει θετικά και θαυμάζω την εισηγήτρια γιατί πραγματικά ε, έδωσε μεγάλη σημασία σε, αυτό, σε αυτή την έκθεση γιατί πολλές φορές ο νομοθέτης ε, κάνει το λάθος να πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να εργαστεί σε βάθος, ιδιαίτερα από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στα κράτη-μέλη. Δώσατε λοιπόν όλη σας την ενέργεια σε αυτή την έκθεση. Σε σχέση με την νομική βάση, το θέμα είναι σαφές, δεν πρέπει να επεκτείνουμε τη νομική βάση. Πιστεύω επίσης ως προς τη μη μεταβιβασιμότητα των αδειών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπε η κυρία Μπερζερό, Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι άνδρες δεν χρησιμοποιούν αυτές τις άδειες εκτός και αν δεν είναι μεταβιβάσιμες. Άρα για να βελτιώσουμε τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν οι άνδρες στη φροντίδα των παιδιών. Έχω υποβάλει τρεις τροπολογίες και μερικές τις ανέφερε η κυρία Μπερζερόν. Καταρχήν η 75. Όταν μιλάμε για ευέλικτες συνθήκες εργασίας και ευέλικτο ωράριο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει καμία διάκριση υπό αυτή την έννοια. Επίσης, η τροπολογία μου 144 μιλά ακριβώς για το ίδιο. Όταν μιλάμε για ευέλικτο ωράριο, Εάν υπάρχουν αποκλήσεις, τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο εργασίας μετά την άδεια. Αυτό απορρέει από τη βασική οδηγία η οποία αναφέρει ότι μετά την άδεια ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ε, επανέλθει στην εργασία ισότιμη εργασία μετά την ε, άδεια, γιατί δεν μπορεί να είναι σίγουρος ή σίγουρη ότι θα έχει την ίδια θέση όπως πριν από την άδεια, αλλά τουλάχιστον να είναι ισότιμη η θέση την οποία θα καταλάβει μετά. Θα πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε και τις ημέρες αδειοδότησης των φροντιστών. Η 122, η τροπολογία μου μιλά για άδεια 12 ημερών από 5 και ίσως θα πρέπει να αποδείξουμε και τις, ε, την ιατρική κατάσταση του φροντιζόμενου. Δεν ξέρω ε, κατά πόσο τα κράτη-μέλη που έχουν ε, εμπειρία μπορούν να μας το καταδείξουν αυτό, αλλά νομίζω ότι πέντε ημέρες είναι λίγες αναφροντιστή κατέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φεραγκούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπερζερόν για την εργασία. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν που θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει τις συνθήκες για να υπάρχει σωστή αντιστήχηση ανδρών γυναικών και ε, συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, έτσι ώστε να υπάρχουν άδειες για τους φροντιστές, να υπάρχει άδεια πατρότητας και γονεϊκή άδεια που να μην είναι μεταβιβάσιμες. Βεβαίως, ε, η άδεια των φροντιστών που ανέρχεται στις πέντε ημέρες είναι πολύ χαμηλή. Το ίδιο αφορά και τις ε, περιπτώσεις ε, ανωτέρας βίας. Το ΕΛΚ έχει υποβάλει τροπολογίες ε, για τη βελτίωση. Βεβαίως για την γονεϊκή άδεια μιλήσαμε για 8 αντί για 12 χρόνια γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την παιδική ηλικία, δηλαδή μέχρι τα 8 χρόνια, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε και τα 12, γιατί θα το διαπραγματευτούμε εάν οι άλλοι θέλουν περισσότερα περισσότερο διάστημα. Επίσης, οι τέσσερις μήνες θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμοι, γιατί φυσικά θα πρέπει να παρέχονται οι περισσότερες φροντίδες σε αυτή την ηλικία. Έχουμε μία καινοτομία μου τροπολογία που μιλάμε για επέκταση αδειών τη στιγμή που υπάρχει αναπηρία. Αλλά κανείς δεν μιλά για μεγαλύτερη άδεια αν η γυναίκα ή ο άνδρας είναι ανάπηρη. Εάν υπάρχει αναπηρία, γονεϊκή αναπηρία, τότε θα πρέπει να αυξηθούν οι άδειες κατά 50% γιατί αυτό έχει σχέση με την ε, μητρότητα και την ε, σεξουαλικότητα των ε, γυναικών που παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας. Γι' αυτό όταν η μητέρα έχει κάποια μορφή αναπηρίας, τα πράγματα δυσχεραίνονται. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή την περίπτωση αναπηρίας των γεννητόρων. Επίσης, εάν υπάρχει εξάρτηση κάποιου τύπου στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα. Ως προς την περίπτωση της κάλυψης εξόδων θα πρέπει να δούμε τι καταβάλει ε, κάθε κράτος ε, για την αναπηρία. Στην Ισπανία καλύπτουμε το 100%, αλλά στη Μάλτα ή την Κύπρο η αναπηρία καλύπτεται λιγότερο. Άρα υπάρχει φυσικά ανισότητα. Προτείνουμε ένα ενιαίο πλαίσιο και θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναπηρία να καλύπτεται κατά το 80% του μισθού για να μην υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ ενός κράτους μέλους και άλλα. Επίσης, θα πρέπει η επιθεώρηση εργασίας να ξαναειδωθεί και να περάσουμε από τα δύο στα τέσσερα χρόνια γιατί από την πείρα που έχουμε βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη μεταφορά του ρυθμιστικού πλαισίου. Υπάρχουν οι οικονομικές προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε στα τέσσερα χρόνια. Εμείς θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες ένα χρόνο, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα άλλα κράτη-μέλη και θα πρέπει να έχουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Και υποβάλαμε και ορισμένες τροπολογίες για την νομική ασφάλεια κατά την περίοδο, τη μεταβατική περίοδο, που θα πρέπει να βελτιωθούν. Εν πάση περιπτώσει έχει σημασία να επέλθει η συμφωνία και η καθήλυν αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει τροπολογίες μέχρι τον Απρίλιο. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε αυτή την πρόταση μέχρι τότε, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ως προς την ισότητα των δύο φύλων και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μπερζεόν γιατί θα μπορέσει να διαπραγματευτεί στη συνέχεια όλα τα θέματα. Ευχαριστώ. ε, ευχαριστούμε πολύ το λόγο. Έχει τώρα ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον διάβασα το σχέδιο νομοδότησης ε, της εισηγητρίας αλλά και η παρουσίαση που έκανε ήταν ε, πάρα πολύ πλούσια. Ουσιαστικά σχολίασε τις περισσότερες από τις τροπολογίες, γι' αυτό και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τη συζήτηση που έχουμε ήδη κάνει. Απλά θέλω να πω στην εισηγήτρια ότι συμφωνώ αρκετά με τη φιλοσοφία τη, δηλαδή ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που υπάρχει στα διάφορα κρατημέλη, προκειμένου να κατατεθεί μια αρκετά ευέλικτη πρόταση, ώστε να μπορεί να γίνει δεκτή παντού. Αυτή είναι μια καλή φιλοσοφία που με εμπνέει και εμένα. Όμως, το πρόβλημα είναι πως έχω την εντύπωση ότι δεν την ακολουθεί πάντα τη φιλοσοφία της η και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά την εναρμόνιση του σχεδί... του... της πατρότητας. Στην αρχική πρόταση υπήρχε αυτή η πρόταση για 10 μέρες ε, τουλάχιστον ε, 12 θέλει η εισηγήτρια. Όμως είναι κάπως ανεδαφικό αυτό στο βαθμό που και η ίδια υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη-μέλη πόρο απέχουμε τις ελάχιστες διάρκειες των 10 ημέρων. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε ε, σταδιακά. 10 ε, και ίσως και παραπάνω ε, είναι λίγο υπερβολικό για τη γονική διαρχικά Αρχικά προτείνει τέσσερις μήνες τουλάχιστον ε, και, αρχι... και πηγαίνει έξι ή και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν έχει νόημα να ε, προσπαθούμε να δούμε τι ισχύει στα κράτη-μέλη αν δεν το λαμβάνουμε υπόψη στη συνέχεια και θέτουμε τελικά υπερβολικά φιλόδοξους στόχους. Νομίζω ότι είναι κακό να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν πολύ ε, βαθιές ρηξικέλευτες αλλαγές στο δικαιό τους. Πάντως, έχω καταθέσει και την τροπή 153 με τη φιλοσοφία της εισηγήτρας που προτείνω το άρθρο 13 ε, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις ε, να γίνει λιγότερο αυστηρό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προβλέπουν σε περίπτωση παραβίαση των δικαιωμάτων εγκυμένων κυρώσεις στα κρατημέλη, αλλά άπαξ και γίνει αυτό, νομίζω ότι δεν είναι και σκόπιμο να αρχίσουμε να παρεθούμε με όλες αυτές τις ε, κυρώσεις που μπορεί να εφαρμόζονται. Ας αφήσουμε στα κράτη-μέλη ε, τη δυνατότητα να προβλέψουν ε, τις κυρώσεις που θεωρούν ότι θα εγγυηθούν το σεβασμό των δικαιωμάτων. Να αφήσουμε λοιπόν κάποια ευελιξία. Πρώτος, ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μαρίνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σκέψεις εντάχει επί του θέματος. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της. Ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και διαθέσιμη για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία μεταξύ κρατών μελών. Το πρώτο ζήτημα που θα ήθελα να τονίσω έχει σχέση με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών το να ενοποιήσουμε συγκεκριμένα καθεστώτα ε, διαφορετικής οικονομικής ε, ευρωστίας όπως την Φιλανδία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Κύπρο ε, δείχνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική ανάπτυξη και ευρωστία αυτών των χωρών. Είναι σαφές ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή ζωή και γι' αυτό, από αυτό απορρέει ένα σύνολο δικαιωμάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των κρατών να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εγώ στη χώρα μου με την παρούσα κυβέρνηση μπορώ να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά αυτό γίνεται με αύξηση των φόρων. Υπάρχει δηλαδή αντίτιμο. Γιατί πολλές φορές γίνεται επανακατανομή ε, εισοδημάτων και δικαιωμάτων για λόγους εκλογοθυρίας. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική ευρωστία κάθε χώρας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, διευρυνθεί το κράτος προνοίας σε όλες τις χώρες, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕΠ κάθε χώρας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει στην ε, Κύπρο, Βουλγαρία ή και Πορτογαλία συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές που ισχύουν στη Φιλανδία γιατί είναι διαφορετική η οικονομική ανάπτυξη της μίας χώρας από την άλλη. Γι' αυτό αυτή η πολιτική θα πρέπει να είναι συνεργατική δηλαδή να λάβει υπόψη ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και δεν μπορεί να επιβάλλει μία καθολικότητα για όλα τα κράτη που διαφέρουν. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση όταν υπάρχουν και ίσες συνθήκες και όροι. Υπάρχει και ένα θέμα καθαρά συντακτικό που έχει σχέση με μία δική μου τροπολογία. Εμείς μιλάμε για εργαζόμενους, εργαζόμενους που εξαρτώνται από μία συγκεκριμένη εργοδοσία και που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Γιατί ε, ε, θα πρέπει να γίνει μία διαφοροποίηση στα πορτογαλικά ε, μεταξύ Εμπρεγκάδου και Τραμπαλιαντόρ. Είναι ένα θέμα που έχει σχέση μόνο με την πορτογαλική μετάφραση. Δηλαδή, όταν λέμε τραμπαλιαντόρες, είναι σαν να λέμε, σαν να μιλάμε για τους εργάτες, για τους προλετάριους, ενώ εμείς μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για εργαζόμενους που λαμβάνουν ένα μισθό στο τέλος του μήνα δεν μπορούμε να του συγχωνεύσουμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το καθεστώς των φροντιστών, διότι ε, είναι πολύ διαφορετικό για το μισθωτό, όπου ο εργοδότης καλύπτει το, τα δύο τρίτα των εξόδων πρόνοιας δεν θα πρέπει να συγχέουμε τις δύο έννοιες που διαφέρουν από τη φύση τους και εξορισμού. Θα πρέπει να μιλάμε για μισθωτούς στα πορτογαλικά, γιατί σε αυτή την περίπτωση η εργοδοσία καλύπτει τα δύο τρίτα των εξόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ταμεία συνταξιοδότησης. Αυτό είναι και ο λόγος της παρέμβασής μου, καθαρά γλωσσικής φύσης. Η κυρία Χαουτάλα. Πολύ σύντομα. Για τον κύριο Μαρίνιο Πίντο, μην ανησυχείτε, γιατί την ε, εφαρμόζουν την πολιτική αυτή τα κρατη όμως το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Επαναλαμβάνω ότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και αυτή η πολιτική εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Το Κοινοβούλιο πάντοτε ήταν στην πρώτη γραμμή για να δει πώ έχει εξελιχθεί η κοινωνία. Ήρθε λοιπόν τώρα η ώρα και οι άνδρες, οι πατέρες να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά δε, τα ποσοστά απασχόληση θα αυξηθούν σίγουρα με την πολιτική αυτή, θα δημιουργηθούν οικονομικέ ευκαιρίε, ε, οικονομική ανάπτυξη και φορολογικά έσοδα. Και αυτό θα αντισταθμίσει δεχόμενε απώλειε. Αυτό είχα να πω. Κύριε Μαρίνιο, σύντομα κι εσείς. Ήθελα να επισύρω την προσοχή σε αυτό, γιατί στην κυβέρνησή μας ε, έχει μειωθεί η εβδομαδιαία εργασία σε 35 ώρες εβδομαδίως, αλλά έχει προβεί σε εκθετική αύξηση των φόρων. Δηλαδή δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό έχει γίνει και για τους έμεσους φόρους. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε το διπλό αντίτιμο για ένα λίτρο ντίζελ. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στο δημόσιο τομέα υπάρχει μείωση της εβδομαδίας εργασίας αλλά διπλασιασμός των πόρων, των, ε, με συγχωρείτε, διπλασιασμός των ε, φόρων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μην γίνονται αυτές οι παραβιάσεις που είναι ανούσιες. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα εκεί που δεν υπάρχει ισότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν, παρακαλώ, πως θα ήθελα να λάβει το λόγο. Ουδής. Α, υπάρχει εκπρόσωπος. Όχι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για εμάς. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που βλέπουμε ότι φαίνεται να υπάρχει βρέα συμφωνία με τους στόχους της πρότασης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους. Διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν μια σύμβαση εργασία ή μια εργασιακή σχέση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και οι μερικώς απασχολούμενοι, οι απασχολούμενοι με συμβάσει ορισμένου χρόνου ή αυτοί που έχουν μια εργασιακή σχέση με μια ε, εργασία προσαρμή απασχόλησης, αλλά όχι τους ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση εργασία ή κάποια εργασιακή σχέση. Αυτό σημαίνει ότι τους γνήσια ανέργους δεν τους περιλαμβάνει. Υπάρχουν ιονοί ε, αυτοαπασχολούμενοι που θα τους ε, εξετάσουμε περίπτωση κατά περίπτωση, αλλά η οδηγία τους ε, αυτοαπασχολούμενους δεν τους περιλαμβάνει. διότι πρέπει να δούμε και τον ορισμό της, ε, του δικαστηρίου για, την, ε, για τον εργαζόμενο. Εκεί δεν ορίζεται ο αυτοαπασχολούμενος. Διορθώνει διεθνές, δεν έγινε λόγος για ανέρους, αλλά για αυτοαπασχολούμενους. Και τώρα ένα σημείο που θέλω να σχολιάσω για την γονική άδεια. Ακούστηκαν κάποια επιχειρήματα για την αύξηση της διάρκειας της γονικής άδειας για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε τη συλλογιστική. Όμως, ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η οδηγία λοιπόν ως έχει δεν προβλέπει μεγαλύτερες ε, περιόδους για τους ε, γονείς με αναπηρία ή για τις μονογονικές οικογένειες κτλ. Διότι αυτό θα σήμαινε ότι οι γυναίκες παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας. Εξάλλου περιοδηγίας πρόκειται, άρα μιλάμε για κατώτατα πρότυπα και δεν εμποδίζει κανείς τα κράτη-μέλη να προβλέψουν ε, μεγαλύτερες περιόδους άδειας εφόσον το θεωρούν απαραίτητο. Το ίδιο ισχύει και για τη διάρκεια, παράδειγμα χάρη για την άδεια των φροντιστών. Είπατε να είναι πιο πολλέ ημέρε. Εμεί αυτό το βλέπουμε σε συνεργασία με τις ευέλικτε ε, ρυθμίσεις ε, της εργασίας ε, για να είναι λιγότερο το βάρος των εργοδοτών αφενός, αλλά κυρίως για να γίνει ένας διακανονισμός για το φροντιστή και προσαρμογή του ωραρίου εργασίας σχετικά με την περίπτωση βέβαια. Μπορεί να μην προβλέπονται, να μην καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις με τις πέντε ημέρες που προβλέπουμε τώρα. Το θέμα είναι να συνδυαστεί οι ανάγκες αυτές ε, με τις ε, ανάγκες ε, για τον φροντιζόμενο και τις ρυθμίσεις. Αυτό θα καλύψει τις ανησυχίες και θα επιτρέψει και στις γυναίκες να μπορούν να εργάζονται πιο γρήγορα. Κυρία Μπερζερό, 27 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 27 Φεβρουαρίου. Κυρία Μπερζερόν, ναι, μένω με την τελευταία φράση της Κομισιόν, ότι ουσιαστικά η επιστροφή των γενικών στην αγορά εργασίας είναι ο στόχος. Όμως, για μένα, το κείμενο γίνεται φιλοσοφικό και ανθρωπολογικό. Μέχρι πρόσφατα οι άνδρες υποτίθεται ότι ήταν αυτοί που εργάζονταν εκτός ε, εστίας και έφερναν τα χρήματα πίσω. Πολλές φορές όμως σήμερα βλέπουμε οι γυναίκες να μείβονται περισσότερο από τους άνδρες. Έχει αλλάξει ε, η εικόνα και αυτό που θέλουμε είναι η σομερή συμμετοχή ανδρών και γυναικών ε, και στην ανατροφή των παιδιών για να καταλάβουν και οι άνδρες, γι' αυτό υπάρχει αυτή η υποχρέωση και για τους άνδρες, ότι έχουν και αυτή η υποχρέωση στην εκπαίδευση στην ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό επανέρχομαι στην ηλικία 8, 13, 12, 14. Νομίζω ότι ο έφηβος βρίσκεται σε μια πολύ ευάλωτη ηλικία και όταν είμαστε 14 ακόμα παιδιά είμαστε ουσιαστικά. Καταλαβαίνω βέβαια ότι και τα μικρά παιδιά ε, χρειάζονται την ε, πλήρη φροντίδα μας, αλλά και η εφηβεία ε, είναι μια δύσκολη ηλικία, θα πρέπει να το δούμε και περνάνε κάποιες εξετάσεις που μπορεί να τους δυσκολεύουν, τους εφήβους είναι σε δύσκολη φάση, θα έπρεπε οι γονείς να μπορούν να περνάνε άδεια. Η Γερμανία δεν δίνουν μια μέρα άδεια, ε, αυτό που είπες. Δεν δίνει καμία άδεια πατρότες. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ενώ η Πορτογαλία, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Μαρίνιο, δίνει 20 μέρες. Άρα η ανισότητα αυτή δεν έχει να κάνει με το οικονομικό σύστημα, αλλά με την φιλοσοφία της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη κατάθεση τροπολογίων και η προποθεσμία που έδωσα προηγουμένω αφορά το επόμενο θέμα που θα καλύψετε πάλι κυρία Μπεζερό εσεί ε, με την τρισδιάστατη εκτύπωση ε, αντικειμένων, οπότε έκανα λάθο. Ε, συγγνώμη, νόμιζα ότι θα ήταν το απόγευμα. Δεν έχω ξαναδιαβάσει το κείμενό μου. Οπότε μπορεί να κάνω λάθη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αυτό το ζήτημα ε, της τρισδιάστατης εκτύπωσης, ε, το καταλάβατε, με απασχολεί πάρα πολύ. Ε, κατά τις συναντήσεις μου γνώρισα πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ε, οι οικονομικές προκλήσεις, ε, αλλά και οι ηθικές και οι νομικές και τα ζητήματα ασφαλείας είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά για την ώρα. Κάποιοι εξημών μπόρεσαν μπορέσατε να ε, επισκεφθείτε τη Ματεριαλή στην επιχείρηση στη Λουβά. Ε, εγώ δεν πήγα, αλλά έχω δει και άλλε τέτοιου είδου επιχειρήσει. Πριν από μερικέ εβδομάδε πήγαμε. Ε, πρωτοστατή στην καινοτομία και την κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων. Σα ενδιέφερε πολύ αυτή η συνάντηση. Πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν γιατί το κανονίσαμε τελευταία στιγμή, αν όμως σας ενδιαφέρει μπορώ να προβλέψω μια νέα συνάντηση στην ε, επιχείρηση αυτή. Προσπάθησα στο σχέδιο έκθεσης να σας κάνω έναν απολογισμό της ε, υφιστάμενης κατάστασης. Κάποια ζητήματα και ερωτήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση επειδή δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σημαντικοί κανόνες για το μέγεθος του κειμένου που πρέπει να σεβαστούμε. Όμως ε, θα ήθελα να τα καλύψω με μελλοντικέ τροπολογίες και μιλάω για την, ανιχνηλασιμότητα, τη ε, κατασκευή τη. της τις εκτύπωση αντικειμένων ε, σε σχέση με τα δικαιώματα του δημιουργού, για παράδειγμα, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, δεν θα θέλαμε να γίνεται παράνομη ε, εκτύπωση προστατευόμενων αρχείων. Ε, νομίζω ότι έχω καλύψει πάντως τις περισσότερες ανησυχίες στο σχέδιο έκθεσής μας ε, κατόπιν της τελευταίας μας συνάντησης για το ζήτημα αυτό. Τα ζητήματα τα ηθικά που αφορούν για παράδειγμα την τρισδιάστατη εκτύπωση στον ιατρικό τομέα και αναφέρομαι στα εμφυτεύματα, τα ζητήματα ασφαλείας ε, για, την, για, τα, για τα όπλα και τους απαραίτητους ελέγχους, όπως επίσης και τα οικονομικά πλεονεκτήματα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα, περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που μπορεί να υπάρξουν από την εκτύπωση αυτή. Δεν πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ αυτός ο κίνδυνος, γιατί δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, πραγματικό πρόβλημα σήμερα. Ε, θα θέλαμε όμως να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί τις συνέπειες για τα δικαιώματα δημιουργών και τη αστική ευθύνης ειδικότερα για την ανάπτυξη της, της διάστατης εκτύπωσης υπάρχουν οι κανόνες και για τα ζητήματα τα ψηφιακά και για τα ζητήματα τεχνικής νοημοσύνης ε, αλλά και για την αστική ευθύνη και την πνευματική διοκτησία. Δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε την καινοτομία με όλο και περισσότερη νομοθεσία αλλά θέλουμε να κάνουμε μία πρόβλεψη και να δούμε κατά πόσο οι υπάρχοντες κανόνες θα πρέπει να γίνουν πιο εξειδικευμένοι ή να προσαρμοστούν. Θα ήθελα τώρα να ακούσω τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, γρήγορη παρουσίαση. κύριος ε, Λουίς Ντεγκράντες Πασκουάλ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητριά για την ε, γενική αυτή ε, έκθεση των ιδεών που σας ενέπνευσαν για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ε, θα είμαι και εγώ σύντομος, αλλά θα σχολιάσω κάποια θέματα που κατά την άποψή μας έχουν να κάνουν ε, περισσότερο με τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες προσφέρει η νέα τεχνολογία. Γιατί αυτή η τρισδιάστατη τεχνολογία δεν είναι επιστημονική φαντασία. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι ήδη υπάρχει. Και μιλάμε για νομικά προστατευόμενα αγαθά. Είναι κάτι ιδιαίτερο σαν καινοτόμο, προσφέρει πλεονεκτήματα. Μειώνει τα γενικά έξοδα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης των προϊόντων. Αυτό είναι προφανές. μπορούν να γίνουν ε, οι πολλαπλές αυτές ε, αντιγραφές του πρωτότυπου πολύ εύκολα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το, σημαντικές οι δυνατότητες οικονομικές και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ εύστοχα. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας με την υφιστάμενη νομική βάση Ιδίω στην ε, περίπτωση των πνευματικών δικαιωμάτων μα καλύπτει, υπάρχουν επαρκή εχέγγυα και ασφαλιστικέ δικλείδες για του εργαζομένους στον τομέα αυτό. Μήπω θα έπρεπε να έχουμε ένα σου εγκαίνερης δικαίωμα για αυτέ τις επιχειρήσεις τρισδιάστατη εκτύπωση, Το νομικό πλαίσιο αρκεί για να καλύψει ε, τις περιπτώσεις ε, τη ευθύνης. Είναι πολλέ ε, οι ερωτήσει ήδη, αλλά υπάρχουν και πολλέ άλλε που θα μπορούσαν να είχα διατυπώσει, γιατί πρόκειται για κάτι καινούριο που γεννά και νέες ευθύνες. Σίγουρα χρειάζεται να πούμε ότι μόλις έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και θα πρέπει να έχει τα κατάλληλους, τους κατάλληλους πολιτικούς κανόνες η Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτό το τόσο πολύπλοκο ε, ζήτημα. Γιατί θα υπάρξουν σίγουρα προβλήματα ή ε, τα πραγματικά δικαιώματα. Πολύ σωστά αναφέρθηκε σε αυτά η, η συγγήτρια. Η, ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρισδιάστατης εκτύπωσης ε, δεν είναι πολλές ακόμη. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί ο αριθμός τους. Πρέπει λοιπόν να ε, βοηθήσουμε ούτε ε, και να μην μειώσουμε, να καταστήλουμε την καινοτομία. Είναι κάρσιο το θέμα και επηρεάζει όχι μόνο τους κανόνες σχεδιασμού, αλλά και τους νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων δημιουργού. Η τρισδιάστατη εκτύπωση λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί, να αξιολογηθεί με βάση όλο το φάσμα ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη της κατηγορίας των προϊόντων. Τα δικαιώματα δημιουργού προστατεύουν την πρωτοτυπία ε, και το δικαίωμα παραγωγής του προϊόντος από τον παραγωγό, από τον δημιουργό. Άρα θα μπορεί σε περίπτωση αντιγραφής ο παραγωγός, ο δημιουργός να ζητήσει αποζημίωση. Ψηφιακό, δίκτυο, ε, ψηφιακό αρχείο συγγνώμη, θα μπορούσε να προστατεύει όπως γίνεται με τα προγράμματα πληροφορικής. Θα ήταν θετικό αυτό, αλλά υπάρχουν ε, ζητήματα, υπάρχουν ερωτήματα. Ένα προϊόν που το σκέφτηκε κάποιος, ε, ψηφιακά το σχεδίσε κάποιος άλλος και το εκτύπωσε ένας τρίτος. Σε ποιον ανήκει το άτομο που σχεδίασε το έργο και αυτός που το ε, σχεδίασε ψηφιακά είναι συνδημιουργή, όπως ορίζει η νομοθεσία περί δικαιωμάτων δημιουργού. Μπορεί να προστατευτεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα ε, προϊόν. Και ποιος είναι ο συνεφευρέτης, ε, ποιος είναι εφευρέτης, υπάρχουν συνεφευρέτες. Είναι πολλά τα πολύ λογικά ερωτήματα απέναντι σε αυτό το καινοτόμο εργαλείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, τύπος προστασίας που θα πρέπει να έχουν οι κάτοχοι αυτών των εκτυπωτών, τρισδιάστατων εκτυπωτών. Αν, αν η η ψηφιοποιημένη εικόνα εκτυπωθεί, ε, αυτό μπορεί να συνιστά, παραδείγματος χάρη, ε, αξιόπινη πράξη. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ διεξοδικά ε, τον αντίκτυπο αυτών των τρισδιάστατων εκτυπώσεων. Η αστική ευθύνη είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Γίνεται μια αναθεώρηση από την Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και ίσως θα ήταν δύσκολο να ορίσουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι θα πρέπει με τους κανόνες, τους νέους, να εντοπίζουμε τους υπευθύνου, χωρίς καμία αμφιβολία. Και να δούμε ο παραγωγός του πληρογράμματος πληροφορικής, η... ο εκτυπωτής, ε, το, το άτομο που χειρίζει τον εκτυπωτή, ο συγκεκριμένος ε, ε, χειριστής, ποιος έχει την ευθύνη τέλος πάντων ε, σε περίπτωση προβλήματος σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του προϊόντος. Το ότι είναι ψηφιακό αυτό το προϊόν σημαίνει ότι μπορούν οι ζητοδιενικέ αυτά πάντα να τροποποιούνται. Τα αρχεία λοιπόν σε ανοιχτό κώδικα θα μπορούν να τροποποιηθούν, να βελτιωθούν και να εξατομικευθούν. Υπάρχουν ερωτήματα ανοιχτά θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε αυτή την πράγματι συναρπαστική τεχνολογία. Αλλά η πρόκλησή μα είναι να δούμε από τώρα ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη εφαρμογή αυτή τη τεχνολογία για το σύνολο τη οικονομία. και τι επιπτώσει θα έχει στην καθημερινή μα ζωή αυτή η τεχνολογία. Αυτέ είναι οι σκέψει μου, κύριε Πρόεδρε. Και φυσικά θέλω να ε, συζητήσουμε, να σκεφτούμε και μαζί με την Κομισιόν να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο που θα ανοίξει την πόρτα και θα ρίξει φως σε έναν ε, νέο κόσμο που πρέπει να τον ε, συνηθίσουμε για να μην μας καταλάβει εξαπίνης ε, η εξέλιξη στον τομέα αυτό. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τεχνολογία της ε, εκτύπωσης τριών διαστάσεων είναι συναρπαστική και καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να συναρπάζει και να ενδιαφέρει και την εισηγήτριά μας. Όμως ε, πρέπει να κρίνουμε μία έκθεση όχι μόνο ως προς το αντικείμενο της μελέτης αλλά και ως προς, το, ε, προς, τις συστάσει ε, που κάνει. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι χρησιμεύει αυτή η έκθεση, γιατί ποια είναι τα νομικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν αυτέ οι νέε τεχνολογίε τρισδιάστατη εκτύπωση. Πρώτο πρόβλημα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι το πρόβλημα τη ε, πνευματική ιδιοκτησία. Το είπε και η ίδια ε, το Ανώτατο Συμβούλιο Ακαδημαϊκής και Λογοτεχνικής Παραγωγής είπε ότι για την ώρα δεν μπορεί να λύσει η τρισδιάστατη εκτύπωση το πρόβλημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, εντάξει, δεν είναι κάτι κατεπήγον, ε, καλό είναι να το σκεφτούμε, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να τρελαθούμε κιόλα. Ε, έχουμε χρόνο να το σκεφτούμε ε, πώς θα κινηθούμε. Το δεύτερο, το δεύτερο πρόβλημα που μπορεί να είναι το πρόβλημα της ευθύνης ε, στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων. Έχουμε την οδηγία μας ε, ε, σχετικά με το θέμα αυτό και λέει η συγγήτρια ότι πρέπει να ισχύει και για τη συγκεκριμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αλήθεια είναι και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει ένα προβληματισμό για το θέμα αυτό, ώστε να υπάρξουν οι ενδεχόμενες διευκρινήσεις αν υπάρχουν ε, αμφιβολίες. Άλλο νομικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ε, ευρύτερης αστικής ευθύνης, ε, γιατί σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν κανόνες γενικής αστικής ευθύνης που καλύπτουν και το πρόβλημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οπότε δεν καταλαβαίνω την πρόταση του σημείου 10 που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τη πιθανότητα δημιουργίας ενός καθεστώτος αστικής ευθύνης ε, δεν, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί δεν χρησιμεύει σε τίποτε αυτή η έκθεση γιατί λέει ότι πρέπει να σκεφτούμε τα νομικά ζητήματα γύρω από το θέμα αλλά έχει ξεκινήσει ήδη αυτός ο προβληματισμός το μόνο που έχει νόημα είναι η τελευταία πρόταση ε, ότι υπάρχει έτσι μία ας πούμε φεντεραλιστική προσέγγιση από πλευράς της ε, εισηγήτριας ότι αυτοί οι νέες τεχνολογίες ε, ε, τρισδιάσταση εκτύπωση. Ε, ε, εκτύπωσης. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί είναι να ε, μπει στα χωράφια έτσι της εθνικής νομοθεσίας και εγώ βλέπω ότι υπάρχει κάτι το πολύ επικίνδυνο εδώ. Θα έπρεπε να μας είχε εξηγήσει για ποιο λόγο θα ήταν προβληματική η διασυνοριακή εφαρμογή αυτή τη τρισδιάστατης εκτύπωση και όχι να μας αναφερθεί μόνο στα εθνικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να, βοηθήσω, να ευχαριστήσω τη Ζωέλ Μπερσογόν, γιατί ε, ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή τη έκθεση γιατί η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένα ε, ζήτημα το οποίο ε, το συζητά πλέον όλος ο κόσμος και είναι λογικό είναι πολύ λογικό και εμείς να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε επί των συνεπειών, ειδικότερα ε, εφόσον οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές αρχίζουν να υπάρχουν πλέον στις ε, αγορές. Ευχαριστούμε και για την οργάνωση αυτής της επίσκεψης στη Λουβά που μας επέτρεψε να δούμε πού ακριβώς έχει φτάσει η εκτύπωση αυτή, τι επιτρέπει, τι δεν επιτρέπει, γιατί υπάρχουν και πολλές ε, ε, φαντασιώσει σε σχέση με το τι κάνει αυτή η εκτύπωση. Ε, συμφωνώ ότι δεν είναι επίγον βεβαίως ε, να αναλάβουμε δράση σε νομοθετικό επίπεδο. Είναι όμως επίγον να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη. Ήταν κατάλαβα καλά, η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ενδιαφέρουσα για την παραγωγή πρωτοτύπων, όμως δεν είναι ενδιαφέρουσα για μαζική παραγωγή γιατί είναι πάρα πολύ δαπανηρή τουλάχιστον για την ώρα. Αυτή η επίσκεψη με βοήθησε μένα πάρα πολύ πάντως. Αυτό που συγκρατώ εγώ από την έκθεση ε, είναι ότι η συγγήτριά μας έχει εντοπίσει δύο βασικά ζητήματα που θα πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, ό,τι αφορά την παραποίηση και την παράνομη παραγωγή, κάτι που δεν είναι καινούριο θέμα, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό. Υπάρχει όμως μια νέα τεχνολογία θα είναι πιο αποδοτική, ε, να δούμε ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε σε αυτήν τη νέα τεχνολογία για να παρεμποδίσουμε την παραποίηση. Και εκεί βέβαια συνδέονται και τα προβλήματα των δικαιωμάτων των δημιουργών, ε, των ευθυνών κλπ. Το θέμα που όλους μας απασχολεί βέβαια πάρα πολύ είναι το θέμα της ασφάλειας των χρηστών, προστασία των καταναλωτών, των παραγωγών κλπ. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι και στην έκθεση να γίνεται η διάκριση μεταξύ της εμπορικής και της ιδιωτικής χρήσης. Γιατί για την εμπορική χρήση νομίζω ότι τα ζητήματα ευθύνης είναι σχετικά προφανή ο παραγωγός είναι υπεύθυνο, ενώ για την ιδιωτική χρήση είναι δική μου η ευθύνη. Αν εγώ παράγω κάτι το οποίο δεν στέκει, για παράδειγμα. Είναι λοιπόν άχρηστο να βλέπουμε τι γίνεται με τους εκτυπωτές δύο διαστάσεων για να δούμε κατά πόσο η νομοθεσία που υπάρχει και τα κριτήρια που υπάρχουν εκεί μπορούν να ισχύσουν και για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Εγώ δεν το έκανα αυτό, δεν έκανα αυτήν τη σύγκριση, δεν έκανα καν την προσπάθεια, σας το ομολογώ, όσον αφορά το δίκαιο του δημιουργού, τα δικαιώματα των δημιουργών. Ε, πάλι το ίδιο ερώτημα τίθεται, πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτά. Υπάρχει μια, ένας κοινός κατάλογος ή όχι, πώς ορίζουμε τα έργα τέχνης, αν υπάρχουν κοινά κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα εξετάσουμε. Επίσης, αναρωτήθηκα για το εξής θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτική χρήση για τους εκτυπωτές που είναι σπίτι τους με τον μικρό τους εκτυπωτή και πάνε σε ένα site ή σε μια πλατφόρμα του ίντερνετ μπορούσε να υπάρχει ένα σήμα ασφαλείας γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο να αντιγράψει κανείς από οποιοδήποτε site κάτι αν όμως υπάρχει μια κάποια εγγύηση θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε την προστασία του ιδιωτικού χρήστη. Νομίζω ότι ο εμπορικός χρήστη του ή άλλω έχει υποχρεώσει που είναι πολύ διαφορετικέ και πολύ υψηλότερο επίπεδο και ισχύουν οι γενικοί κανόνε εκεί. Ο φόβο λοιπόν τη παραγωγή επικίνδυνων ε, προϊόντων είναι θεμητός νομίζω, όμως δεν ε, ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτό. Αυτό παραμένει ένα ένας παράγων ανησυχίας, αλλά νομίζω ότι πέρα από όλες τις ανησυχίες ε, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ε, τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής που είναι συναρπαστική, που ανοίγει προοπτικές ε, για τις χώρες μας. Για κάποια νέα παραγωγή ενδεχομένως σε κάποιες χώρες, σε κάποιες χώρες ε, οι χώρες βέβαια που θα μπορούσαν να φέρουν το κόστος ε, αυτής της ε, παραγωγής θα μπορούσε αυτό λοιπόν να έχει ένα εποφελές αποτέλεσμα ακόμα και στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τούτου λεχθέντος βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό και με πολύ χαρά εγώ θα συνεισφέρω ε, αν όχι στη βελτίωση, τουλάχιστον στην ε, ε, διαφώτιση κάποιων στοιχείων που αναφέρθηκαν σήμερα. Θα πρέπει να αποφύγουμε το τέλεαρ να μιλήσουμε για άλλες διαστάσεις του προβλήματος εκτός από τις νομικές. Εδώ συμφωνώ με τον κύριο Λεμπρετών ότι έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό προβλημάτων που μας απασχολούν. Ε, και ίσως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός ε, νομικών προβλημάτων, αλλά και αυτό είναι εκτιμητέο. Μαρίνιο Πίντου. Ευχαριστώ εντάχει. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στις σκέψεις του κυρίου Λουίς Γκράντες που σχετίζονται με αυτή την τεχνολογία εχμής. Επίσης ένα θέμα καθαρά γλωσσικό. Εγώ ήμουνα ένας από τους λίγους ευρωβουλευτές που επισκέφτηκα αυτή την επιχείρηση τρισδιάστατης παραγωγής. Και ε, έλαβα υπόψη την όλη διεργασία και διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, ότι αυτή η νέα τεχνολογία δεν έχει να κάνει με την εκτύπωση. Ε, αφορά ένα λογισμικό που εισάγεται. Αυτό θα έχει επιπτώσεις ε, μεγάλη σημασίας, ζωτική σημασίας. και εμείς θα πρέπει να προβλέψουμε να προβλέψουμε αυτές τις ε, εξελίξεις για να ε, θεραπεύσουμε ή να προβλέψουμε. Γιατί με έναν τέτοιο εκτυπωτή, τρισδιάστατο εκτυπωτή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, μπορεί να γίνει και κακόβουλη χρήση, παραδείγματος χάρη στον τομέα της ε, κατασκευής όπλων όπου ε, έγινε χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή για περίπτωση, σε περίπτωση οπλοχρησίας, όπως είδαμε από την τελευταία είδηση της μαφίας που χρησιμοποίησε αυτή την τεχνική για να φτάσει και στη δολοφονία. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ολέθριες συνέπειες που ενδεχομένως θα είχε και η χρήση αυτής της τεχνολογίας. θα πρέπει να περιοριστούμε στα νομικά θέματα. Άντερσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το εκπληκτικό θέμα. Αυτή η τρισδιάστατη εκτύπωση εξελίσσεται δραστικά και ίσως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διδάσκεται και στα σχολεία, όπως ισχύει στην περίπτωση της ε, Σουηδίας, ενός σχολείου στη Σουηδία. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο σύστημα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πρωτότυπα και έτσι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε νέες τεχνολογίες δημιουργώντας και εξαρτήματα και θα μπορούσε να είναι και μέσον καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που με βρίσκουν σύμφωνο σε αυτή την έκθεση, αλλά δεν θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να συρρυκνώσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία. Και δεν θα πρέπει να πλήξουμε αυτή την τρισδιάστατη τεχνολογία. Και θα πρέπει να, σας, να μας απασχολήσουν ορισμένες πτυχές αυτής της έκθεσης. Υπάρχουν στοιχεία που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσουν. Ας αρχίσουμε από το γλωσσικό. Αλλά ίσως υπάρχει και θέμα μετάφρασης. Στο γιώτα όπου γίνεται λόγος για τρισδιάστατες εκτυπώσεις ε, και ενώ όλες δεν είναι παράνομες, μερικές θα μπορούσαν και να είναι. Δεν ήταν αυτός ο, ίσως ο στόχος, δεν ήταν ευτυχής αυτή η διατύπωση. Επίσης, δεν ε, έχουμε, δεν γίνεται μνήα στη δυσδιάστατη εκτύπωση. Έχουμε ήδη εκτυπωτές που είναι πάρα πολύ καλοί και ακριβείς ως προς τις δυσδιάστατες εκτυπώσεις. Αλλά δεν έχουμε ένα διεθνές σύστημα εποπτείας έτσι ώστε να μην γίνουν εκτυπώσεις ή να τυπωθεί υλικό το οποίο αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει θέμα και όταν κατεβάζουμε υλικό στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, ε, μουσική ή ταινίες. Θα μπορούσε ε, λοιπόν να εισαχθεί ένας αριθμός, μέγιστος αριθμός τρισδιάστατων εκτυπώσεων ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ιδιωτική χρήση. Επίσης, ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε ένα φόρο για τις ε, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, αλλά δεν μπορεί να εισαχθεί ένας φόρος για κάθε χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας περιορισμός, νομίζω, ακόμα και λεκτικός. Επίσης υπάρχουν θέματα ως προς την ευθύνη και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι και να προλάβουμε το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι το θέμα που προανέφερε ο συνάδελφος είναι μεγάλο, έχει μεγάλες διαστάσεις, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει πρόβλημα ούτε στο μέλλον. Δηλαδή να μην ανησυχούμε αλλά να προλαμβάνουμε. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες σε αυτή την έκθεση και προσβλέπω σε μία εις βάθος συζήτηση. Είναι μια πολύ καλή έκθεση, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοδομητική έκθεση. Ε, χαιρόμαστε που εξετάζετε ενδελεχώς το θέμα και εδώ μιλώ από πλευράς διανοητικής ιδιοκτησίας. Συμφωνούμε με τα συμπεράσματά σας και θα αναλάβουμε δράση. Όπως προαναφέρθηκε από την εισηγήτρια, η υπάρχουν ανησυχίες και ανασφάλεια σε σχέση με την, το νομικό πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε μία μελέτη συλλογή στοιχείων για να δούμε κατά πόσο χρειάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας για να λάβουμε υπόψη πλήρως την τεχνολογία αυτή. Η εργασία αυτή θα αρχίσει το Μάρτιο και θα είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο, αν όλα πάνε καλά. Επίσης ε, έγινε λόγος για ενίσχυση της θετικής πλευράς του, της τρισδιάστατης εκτύπωσης που χρησιμοποιείται από ιδιώτες ή επιμέρους χρήστες και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προωθήσουν τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις και κατά πόσο μπορεί να υπάρχει πιο επικοδομητική χρήση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση αυτών των προτύπων. Επίσης, άκουσα με ενδιαφέρον ενδιαφέρον το θέμα της ανιχνευσιμότητας, όπως είπε η συγγήτρια. Αυτό μας απασχολεί και φυσικά αυτή η χνηλασία είναι πολύ σημαντική και για τη τρισδιάστατη εκτύπωση. Ευχαριστούμε πολύ και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των εργασιών σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλετε κυρία Μπεριζερό ε, να δευτερολογήσετε. Ναι, για δύο δευτερόλεπτα. Για να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο. Νομίζω ότι όλοι με τις διαφορετικές του ευαισθησίες διέκριναν το πρόβλημα. Ο κύριος Ντεγκράντες ε, πολύ καλά τοποθέτησε το ζήτημα και είπε ότι πραγματικά είναι μια ενδιαφέρουσα νέα τεχνολογία που δεν πρέπει να την ε, πάρουμε στα ελαφρά και ο βιομηχανικός κόσμος θα μπορούσε να ε, ωφεληθεί και τα κράτη-μέλη. Αν υπάρχει βιομηχανική παραγωγή, όλα τα εξαρτήματα ε, που παράγει μια επιχείρηση όπως η Ντάρτη, για παράδειγμα, αν ας πούμε πάτε να αλλάξετε ένα κουμπί που έχει σπάσει στο φούρνο, δεν ε, θα πάνε στο εργοστάσιο να το παραγγείλουν, να μπορούν ε, στο πίσω μέρος ε, του καταστήματος να το φτιάξουν αμέσως με τη χρήση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Δεν είναι λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Άντερσον, ένα όνειρο η τρισδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχει από τη δεκαετία του 80, θα αλλάξει την τεχνολογία για πολλά πράγματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ιδιώτες, πολύ σωστά, αλλά χρειάζεται και η χνηλασιμότητα, γιατί τα αρχεία αυτών των ε, εργαστηρίων ε, είναι διαθέσιμα εκατομμύρια σχεδόν. Ε, δεν ξέρουμε ποιος τα έχει βάλει στο διαδίκτυο. Γενικά είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Και δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Και είσαι και νομικός. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε από νομική πλευρά το πρόβλημα αυτό με το πρόσημο ότι δεν έχουμε πρόβλημα μέχρι στιγμής και ε, υπάρχουν ε, ε, τα κείμενα όπως το 1384 για την αστική ευθύνη κτλ. Όχι, είναι μια ειδική τεχνολογία και το καθήκον μας ως νομοθετών είναι να προβλέψουμε τι πρέπει να νομοθετήσουμε. Όλοι σας λοιπόν φωτίσατε διαφορετικές πτυχές και νομίζω ότι καλό θα ήταν να συναντηθούμε από κοινού, γιατί έχουμε σωστά ε, συλλάβει το πρόβλημα, αλλά πρέπει να λύσουμε τα, τις πτυχές των προβλημάτων. Προθεσμία κατάθεσης, λέει ο Πρόεδρος, 27 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Μπορούμε λοιπόν εδώ να κλείσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο σημείο 6 που είναι ο πίνακα αποτελεσμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη δικαιοσύνη του 2017, εξέταση του σχεδίου έκθεση. Η κυρία Γιούτελαντ, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία σε απάντηση στην ε, δημοσίευση του 2017 της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπή για τον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα τη δικαιοσύνη. Τον Απρίλιο συγκεκριμένα του 2017 δημοσιοποιήθηκε αυτό το έγγραφο και μας ε, δίνει μια επισκόπηση ό,τι αφορά την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως μια διαφορά από τις προηγούμενες εκδοχές υπό την έννοια ότι η συγκεκριμένη έκθεση βλέπει και την πρόσβαση των ε, πελατών στη δικαιοσύνη όταν καταφέρονται εναντίον εταιριών και δείχνει επίσης πόσο μακροχρόνιες είναι οι δικαστικές δικασίες σε ό,τι αφορά δικήματα νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης τα ειδικά μέσα, η δίκαιη, η δίκη, ε, όλα αυτά είναι σημαντικές προϋποθέσεις για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ωστόσο, μας δείχνει η εμπειρία μας ότι δεν υπάρχει επαρκής δικαιοσύνη στο δικαστικό σύστημα των κρατών μελών, από τους πολίτες του εκάστοτε κράτους μέλους είναι ε, οι πολλοί μηχανισμοί και παράμετροι που επηρεάζουν ε, το βαθμό εμπιστοσύνης, ό,τι αφορά δηλαδή την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι τόσο σημαντικός. Έγινε μια συνεδρίαση σκηνοδών εισηγητών λίγο πριν ε, σας διαβιβάσω το σχέδιο έκθεση. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική αυτή συνάντηση και χαίρομαι γιατί δείχνει να υπάρχει ευρύ υποστήριξη συνολικά προς την έκθεσή μου. Στο σχέδιο έκθεσής μου λοιπόν καλωσορίζω τον πίνακα αποτελεσμάτων για το 2017 και τους στόχους του, δηλαδή για μια αποτελεσματική ανεξάρτητη ε, δικαιοσύνη ε, και για ε, ποιοτικό δικαστικό σύστημα στα κράτη-μέλη. Όμως, για να κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση και άλλων ε, πηγών πληροφοριών πέραν του πίνακα αποτελεσματών όπως ε, από το Ινστιτούτο Νομικών Μεταρρυθμίσεων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, το Συμβουλίο της Ευρώπης. και ένα από τα θεματικά τμήματα του Κοινοβουλίου. Επίσης θέλω να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου, τονίζοντας την ανάγκη έντασης και διαφοροποίησης των, της εκπαίδευσης των δικαστών για να ενημερωθούν για τη διάσταση του φύλου. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων που επιμένει δυστυχώς. Ιδίω δε ε, στα Στου βαθμού της δικαιοσύνη του υψηλότερου ε, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο βλέπουμε ανισορροπία μεταξύ των δικαστών σε ό,τι αφορά δηλαδή, την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για LGBTI επίσης είναι ένα θέμα. Πρόσβαση στην ε, ε, νομική συνδρομή. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις διάκρισης ή την αντιστροφή του βάρους απόδειξη. Αυτά τα στήματα πρέπει να τα προσέξουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να θαρρύνουμε την Κομισιόν να αναπτύξει συγκεκριμένους δείκτες για να αναβαθμίσει και να προωθήσει τις βασικές αξίες ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων, ε, κράτους δικαίου και στον τομέα τη δικαιοσύνη. Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στην ε, περαιτέρω χρήση των τεχνολογιών ε, πληροφοριών και επικοινωνία στα δικαστικά του συστήματα για να γίνουν πιο προσβάσιμα και κατανοητά από του πολίτε, ακόμη και από αυτού που έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρία. Πιστεύω επίση πω θα ήταν σκόπιμο να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και τι διαδικασίε των συλλογικών προσφυγών ε, στο πρόγραμμα που έχει του χρόνου για την προσβασιμότητα και η Γιούρη σύντομα θα έχει και ε, μάλλον θα έχει ε, στη συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης μια ακρόαση για τους μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας, εξέλιξης και μελλοντικά βήματα. Είμαστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι και καλό θα ήταν να δούμε πώς έχουν τα τρέχοντα συστήματα και οι διαδικασίες ισχύουσες ε, στα κράτη-μέλη, πάντοτε και σε συνάρτηση με του στόχου του πίνακα αποτελεσμάτων. Υπάρχει επίσης ένα χάσμα δεδομένων. Δεν έχουμε δεδομένα από κάποια κράτη-μέλη για συγκεκριμένε κατηγορίες, όπως αναφέρει στον πίνακα αποτελεσμάτων. Προτείνω λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη αυτά να συνεργαστούν πλήρως με την Κομίσιο για να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα τους. Επίσης προτείνω να απευθύνουμε και στα κράτη-μέλη να αποδώσω μεγαλύτερη προσοχή στο γεγονό ότι η ισχυρή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη βασίζεται αφενό στην έλλειψη παρεμβάσεων πιέσεων ε, από πολιτική και κυβερνήσει και από την άλλη στα απαραίτητα εχέγγυα ε, που παρέχει πολιτεία. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει αυτή την έκθεση να τη χρησιμοποιήσουμε για να επωνυδίσουμε κανένα. Γι' αυτό και απέφυγα επιμελώς να αναφερθώ σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Σε ό,τι δεν αφορά το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 6η Μαρτίου. Και στις επόμενες συνεδριάσεις, 26-27 Μαρτίου, θα εξετάσουμε αυτές τις τροπολογίες για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γιούρη 24 Απριλίου, όπως προβλέπετε. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Any member... ε, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θέλει το λόγο, κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Γιωτελάντ. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί εκ του σύνεγγης τις εξελίξεις των πίνακα αποτελεσμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ε, σύστημα δικαιοδοσίας έχει μεγάλη σημασία εδώ και υπάρχει μία συνδεσιμότητα ε, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και μία ε, οικονομία η οποία ανθίζει. Θα υποβάλω μία τροπολογία για να ε, επεκταθούν ορισμένες παρατηρήσεις σε ε, χώρες που έχουν ε, συνθήκες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με, ένα, με τη χρήση ενός ποιοτικού δικαιοδοτικού συστήματος. Μιλήσατε βεβαίως και για το ε, χάσμα των δύο φύλων στα συστήματα δικαιοσύνης ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σκόπιμο. Επίσης, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει μεγάλη σημασία γιατί υπάρχουν ε, χάσματα στη χρήση των ένδικων μέσων. Πολλές φορές οι πολίτες αντιμετωπίζουν προσκόμματα τη στιγμή που γίνεται λόγος για πρόσβαση στον τομέα δικαιοσύνης ε, και τη χρήση δικαστικής αρρωγής. Η έκθεση, η αυτή έκθεση ασχολείται με το ε, εμπορικό δίκαιο το, και το διοικητικό κυρίως, και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να σταθούμε σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια σύγκριση και του διοικητικού δικαίου μεταξύ κρατών μελών για να ε, ασχοληθούμε και με αυτή την πτυχή του θέματος. Θα υποβάλω μερικές τροπολογίες και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε. Στην παράγραφο 10 μιλάτε για την ε, διαδικασία ε, συλλογικής για το θέμα της ένδικης προστασίας και γι' αυτό θα το δούμε και αυτό μέσα στα πλαίσια της ε, μελλοντικής ε, διαδικασίας, του χρόνου δηλαδή, για, ως προς το θέμα της ε, δικαστικής προσφυγής και της χρήσης ένδικων μέσων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρανιέφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Γκούτελαντ για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Βεβαίως, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ε, έχει μεγάλη σημασία, είναι ζωτικής ε, σημασίας για το κράτος δικαίου και για τις δίκες ε, δίκες. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που θα πρέπει ίσως να τροποποιηθούν κάπως. ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή τη χρήση ένδικων μέσων για τη συγκριτική μελέτη για του χρόνου. Σε σχέση με την προσβασιμότητα στα ένδικα μέσα, δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό θα έδινε αντιπροσωπευτικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο 2 μιλάμε για ε, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ΛΟΑΔ. Νομίζω ότι αυτό κάθε αυτό αποτελεί μία διάκριση. Νομίζω ότι η προστασία δεδομένων απαγορεύει την ε, επεξεργασία στοιχείων σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των πολιτών. Θεωρούμε ότι αυτό το βαθμολόγιο θα μπορέσει να αποτιμήσει τα δικαστικά συστήματα, τα συστήματα δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορούμε να, ε, χρησιμοποιήσουμε μόνο στατιστικά στοιχεία. Μαρίνιου Πίντου. Ήδη έχω εκφράσει ορισμένες σκέψεις ε, που θα επαναλάβω. Η δικαιοσύνη είναι ένα αγαθό απαράμιλο το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε στα χέρια των δικηγόρων και των δικαστών. Η δικαιοσύνη είναι ύψης της σημασίας για τις επιχειρήσεις και την οικονομία, όπως είπε και η Χάιντι Χαουτάλα, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες, για την προάσπιση και των δικαιωμάτων των πολιτών και την υπεράσπιση των πολιτών, καθώς και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Υπό αυτή την έννοια ασχοληθήκαμε με τα διάφορα συστήματα δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολλά χάσματα. Υπάρχουν χώρες όπου η δικαιοσύνη αποτελεί ε, ένα είδος ιερουργίας. Είναι υπεράνω όλων. Στη χώρα μου Ε, πρέπει να αποτανθεί κανείς σε έναν ε, δικαστή στη χώρα μου, όπως ε, στα αρχαία χρόνια ένας δουλοπάρικος απευθυνόταν σε έναν πολίτη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία απτή πραγματικότητα. Εάν ένας πολίτης κατά τη Γαλλική Επανάσταση ε, είχε ε, πεθάνει και μπορούσε να αναστηθεί στη δική μας εποχή όπου υπάρχει διαδίκτυο, γυναίκες με ε, μινιφούστες, μία νέα συγκεκριμένη πραγματικότητα. Αυτό θα τον άφηνε έκθαμβο. Όμως, σε ένα δικαστήριο θα έβλεπε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από που, τον καιρό που πραγματικά έζησε. Έχουμε λοιπόν την ίδια ακόμα και ενδυματολογία στα δικαστήρια. Και ο λόγος είναι ίδιος. Η δικαιοσύνη στη χώρα μου δεν έχει αλλάξει και δεν προσαρμόστηκε στις σύγχρονες ανάγκες. Οι γυναίκες μπόρεσαν να γίνουν δικαστές μόνο μετά την Επανάσταση της 25ης Απριλίου. Δηλαδή μετά τη δεκαετία του 70. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν χώρες που είναι παρεμβατικές ως προς τη δικαιοσύνη, που δεν δέχονται τον διαχωρισμό των εξουσιών. Δηλαδή, υπάρχει μία πολιτική ατζέντα που διέπει το δικαστικό σώμα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνομία η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Βλέπουμε ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις οδηγούν σε ασφυξία τον δικαιοδοτικό τομέα και στην Ισπανία ε, το δικαστικό, η δικαιοδοσία μάλλον, το σύστημα δικαιοδοσίας οδηγεί σε φυλακή ανθρώπους που έχουν διαφορετικές πολιτικές ε, πεπιθήσεις. Άρα δεν υπάρχει ε, ίση αντιμετώπιση της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη. Αυτό το αναφέρω είναι γιατί οι δικαστές δεν είναι θεότητες. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο ισχύει και λειτουργεί εξ δέους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη διάσταση του ζητηματός θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δύσκολη προσβασιμότητα στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα ε, απαγορευτικό κόστος και είναι γνωστή η υπόθεση ενός δημοσιογράφου και μιας δημοσίας υπαλλήλου που δεν έκαναν αγωγή για διαζύγιο γιατί δεν μπορούσαν να επομιστούν το κόστος. Και συνεπώς βλέπουμε ότι σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα οι γυναίκες είναι, βρίσκονται πιο μακριά. Και αυτό το βλέπουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τη στιγμή που λέμε ότι τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να ανοίξουν στις γυναίκες, εμείς φέρνουμε το αντίθετο παράδειγμα γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο ούτε στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο, ούτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το μέλλον. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομα. Εγώ θα ήθελα απλώς να τονίσω όλα όσα υπόθηκαν και από τον συνάδελφο Μαρίνιο Ντεπίντου. Ε, σε σχέση με την ισότητα των φίλων ε, και το ε, δικαστήριο. Όλα αυτά πολύ ορθώς υπόθηκαν. Το θέμα που με απασχολεί εμένα είναι ο πίνακας δικαιοσύνης. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα θέσατε ήδη και αυτό αποδεικνύει πόσο πολύ χρειαζόμαστε τον πίνακα αυτό δικαιοσύνης γιατί αφορά την εμπιστοσύνη στα νομικά μας συστήματα. Ένα μόνο θα ήθελα να προσθέσω που πάντοτε ο Λουίτζι Μπερλιγκέρ το έθετε μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση ότι και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει περαιτέρω εκπαίδευση και διαβίου μάθηση όλων των νομικών επαγγελματιών. Γιατί όταν πρόκειται για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη συγκρισιμότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Χρειαζόμαστε εκείνους που ασκούν το επάγγελμα αυτό της δικαιοσύνης και που πολλές φορές ε, τόσο πολύ εστιάζονται μόνο στα εθνικά συστήματα να συμμετέχουν. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να το συμπεριλάβετε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμπρετών. Merci, Ευχαριστώ ε, πραγματικά ε, η έκθεση αυτή επικεντρώνει την προσοχή μας στον πίνακα δικαιοσύνης που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ κρατών γιατί περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία των δικαστών στα κράτη-μέλη. Η έκθεση ενθαρρύνει τα κράτη να ε, επενδύσουν περισσότερα στην εκπαίδευση και βεβαίως ε, μας βρίσκει σύμφωνος αυτός ο στόχος. Για το γενικό στόχο λοιπόν της έκθεσης συμφωνώ. Όταν διαβάζουμε όμως ε, την έκθεση ε, υπάρχει μια μηχανία για ορισμένε πτυχές. Πρώτον, όταν θέλουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν περισσότερο δεν πρέπει να επιμένουμε τόσο πολύ στο γεγονός ότι κάποια είναι σε μειονεκτική θέση ή δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να τονίζουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων ότι υπάρχει το εργαλείο και πρέπει να το ενισχύσουμε και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επιτείνουν τις προσπάθειες προσπάθειές αλλά δεν χρειάζεται τόσο συχνά να, ε, να, να επισημαίνουμε ότι κάποια κράτη δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά. Δεύτερον, είναι λίγο παράξενη η διατύπωση. Στο 11 λέμε για καταναλωτές. Μπορεί να είναι ένα ζήτημα μετάφρασης, αλλά όταν κάποιος ζητά δικαστική βοήθεια δεν είναι πια ε, καταναλωτής, είναι ένας διάδικος. Συνεπώς, δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα. Εμείς ως ευρωβουλευτές πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας διάδικος είναι ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με τον καταναλωτή καταναλωτή. Πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα με εσά, κύριοι συνάδελφοι. Είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και εγώ είμαι ευαίσθητο όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων. Όμω πιστεύω ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε από του δικαστέ να καταπολεμήσουν όλε τι μορφέ διάκριση. Δεν θέλω να τονίσω τη μία μορφή περισσότερο από την άλλη και σε αυτή την έκθεση. Μα εκπλήσει το γεγονό ότι επιμένουμε πάρα πολύ στι διακρίσει σε σχέση με, τους, με το σεξουαλικό προσανατολισμό, με τους ε, ε, ΛΟΑΤ ε, και έχω λίγο κουραστεί με όλα αυτά τα κείμενα που τονίζουν τόσο πολύ αυτή τη διάσταση. Νομίζω ότι καταντά αντιπαραγωγικό και νομίζω ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι ένα σύνολο και πρέπει να καλέσουμε για την, να κάνουμε έκκληση για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων χωρίς να τονίζουμε μία και περισσότερο από τις άλλες γιατί τελικά καταλήγουμε να ε, δημιουργούμε αμφιβολίες για τη σοβαρότητα των διακρίσεων ε, που μπορεί να πλήττουν άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την τελευταία, με την τελευταία παρατήρηση του κυρίου ε, Λεμπρετών. Κύριε Χάουταλα, Προφανώς ο η εισηγήτρια θα μπορούσε να μας εξηγήσει αν ε, υπάρχουν ε, σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι άνθρωποι αυτή της ομάδας ε, ΛΟΑΤ έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα με την πρόσβαση, τη δικαιοσύνη και την νομική αρρωγή. Θα με ενδιέφερε να μάθω κατά πόσο αυτό ήταν ο λόγος που συμπεριλάβατε αυτό το σημείο στην παράγραφο 12 στο σχέδιο έκθεσης. Εγώ θα έλεγα ότι άλλες ευάλωτες ομάδες και μειονότητες ε, θα μπορούσαν και εκείνες να έχουν προβλήματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στη νομική αρρωγή. Από τη στιγμή που συζητούμε λοιπόν την, τον πίνακα δικαιοσύνης που κατήρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, και από τη στιγμή που τροφοδοτείται από πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, θα έπρεπε πιο διεξοδικά να αναφερόμαστε στις ομάδες μειονοτήτων που θα έπρεπε να καλύπτονται από ε, την νομοθεσία μας περί καταπολέμησης των διακρίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Πολύ σύντομα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ σύντομα. Και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την έκθεσή της, ε, τη συναρπιστική και για την επικοδομητική συζήτηση τη σημερινή. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, να βοηθήσουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα δικαστικά τους συστήματα. Πολύ σωστά, το λέει και έκθεση. Τα εθνικά δικαστήρια είναι και ενωσιακά δικαστήρια. Όλοι λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον να είναι καλύτερη, ε, να είναι πιο αποτελεσματικά αυτόνομα και ανεξάρτητα. Έχουμε σημειώσει λοιπόν όλα τα σημεία τα οποία αναφερθήκατε, σας τα αναφερθήκατε σήμερα. Ευχαριστώ. Κυρία Χουγιούτελ, αν θέλει κάτι να προσθέσει. Πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συζήτηση αυτή και τα επικοδομητικά ερωτήματα και σχόλια. Χαίρομαι και εγώ γιατί βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη προς την έκθεση και τα βασικά θέματα. Όπως είπε και η Κομισιόν, πρέπει, είναι σημαντικό και εμείς να βοηθήσουμε την, τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα δικαστικά τους συστήματα και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όπως τα βλέπουμε εμείς, αυτό το πρόβλημα με τα δεδομένα που είπα, που είναι λυπή και άλλα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση, η πιο έντονη διάσταση του φύλου, ανεξάρτητα ισχυρά δικαστικά συστήματα και τους Μαρίνιου Πίντου είπε πολύ εμπνευσμένα λόγια για το θέμα αυτό και άλλοι συνάδελφοι επίσης μίλησαν για τροπολογίες ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε κάποια θέματα. Πολύ ενδιαφέρον θα περιμένω τις τροπολογίες και τη διατύπωση που είπατε εσείς ε, κύριε Λεμπερτών θα το κοιτάξω και αυτό σε ό,τι αφορά τα δύο ζητήματα για τα οποία εκφράστηκαν ανησυχίες. Νομίζω ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων έχει επικριθεί ότι δεν είναι αρκετά συναφής. Ε, δεν περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που θα έπρεπε. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δηλαδή έπρεπε να περιλαμβάνονται και βέβαια ένα από αυτά είναι και τα δικαιώματα των LGBTI συμπολιτών μας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θέλω να επεκταθεί ο πίνακα του να καλύψει και αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς συλλογικής ένδειξης προστασίας. Νομίζω ότι μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε δικαστικές διαμάχες στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε να προσθεθεί και αυτό στον πίνακα αποτελεσμάτων, αλλά θα περιμένω να ακούσω περαιτέρω σχόλια για να δούμε τελικά και πώς θα ψηφίσουμε στο τέλος. Okay. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είπα ήδη ποια είναι, μάλλον υπόθηκε ήδη ποια είναι η προθεσμία κατάθεση τροπλήγων 6 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Είμαστε στην ώρα μας. Ακριβώς.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 Dear ήρθατε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Ε, το θέμα είναι ε, η συλλογική ένδικη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίξεις και μελλοντικά βήματα. Είναι μεγάλη χαρά που ήμουν εδώ ε, μαζί μας εξέχοντες επιρρογνώμονες είμαι βέβαιος ότι, ο, ότι είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ακρόαση σε σχέση με τις πρόσφατες, την πρόσφατη δημοσίευση ε, της εφαρμογής ε, των συστάσεων του 2013 για, την, ε, ε, για τους μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας από το δικαστήριο. Αυτές οι συστάσεις του 2013 δημιουργούσαν κάποιες αρχές σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων ε, υπό το ενωσιακό δίκαιο σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε σχέση και με τα, ε, και με την, ε, και με τα ασφαλιστικά μέτρα αλλά και με την αποζημίωση. Προκύπτει από τη σύσταση ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν συστήματα τέτοιας προστασίας στο σύστημά τους που θα συνάδουν με τις βασικές αρχές χές Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβανομένων υπόψη των νομικών παραδόσεών τους και ε, της εξασφάλισης ε, της μη κατάχρησης. Σύμφωνα με την παράγραφο 41 ε, της σύσταση, πρέπει να, να βασίσει την αξιολόγησή σε βάση της εμπειρίας που έχει για τον αντίκτυπο στην πρόσβαση ε, στη δικαιοσύνη, το δικαίωμα της αποζημίωσης, ε, της παρεμπόδιση καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και της ε, ε, λειτουργίας ε, της ενιαία αγοράς σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα τη Οικονομία τη Ένωση και τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο τα μέτρα ενίσχυσης της οριζόντια προσέγγισης των συστάσεων πρέπει να ε, προταθούν. Θα ήθελα χωρί περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον πρώτο, πρώτο, πρώτο μιλητή μα τον Γιάτσεκ Γκάρξκα, το, το λόγο και μετά ε, στον κύριο Γιώργο από την ε, Γενική Διεύθυνση Just. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας, συνάδελφοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρακτική εφαρμογή των συστάσεων του 2013 ε, προς στην Επιτροπή σας. Ε, πάντοτε εκτιμούμε το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας στις συλλογικές αγωγές, στα συλλογικά, συλλογική ένδικη προστασία για τις συστάσεις ε, που δημοσιεύσαμε ε, το 2013. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε πολλά έτη προηγούμενης εργασίας, κυρίως στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών ε, και του δικαίου ανταγωνισμού. Η σύσταση έχει αυτήν την τεράστια αξία του να αναφέρει ευθαρσός ότι τα, ε, η συλλογική ένδικη προστασία είναι ένας από τους σωστούς ε, τρόπους ε, επιβολής των άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αυτή τη θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε κάποια, κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες προκειμένου να προστατεύσει τη δικαιοσύνη της ε, ε, συλλογικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει την πρακτική εφαρμογή της σύστασης αυτής και η έκθεση η οποία εγκρίθηκε στις 25 ε, Ιανουαρίου του τρέχοντος ε, προβαίνει στην αξιολόγηση αυτή. Πρέπει να τονιστεί ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία της, ε, έκθεση, της έγκρισης έκθεσης ε, συνέπεσε με κάποια γεγονότα τα οποία φάνηκε να είναι πολύ σχετικά ε, με την συλλογική ένδικη προστασία και αναφέρομαι ειδικότερα στο σκάνδαλο για τις εκπομπές αερίων από τα αυτοκινούμενα οχήματα τα οποία δημιούργησαν μια κατάσταση μαζικής ζημίας άνευ προηγουμένου μεταξύ καταναλωτών και επενδυτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα βεβαίως να δούμε ε, πώς ο μηχανισμός αυτός λογικής ένδικης προστασίας λειτουργήσε στα διάφορα κράτη-μέλη. Ένα ακόμη σημείο, ε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την ε, έκθεση αυτή, είναι ε, το αυξανόμενο και ολοένα αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι διασυνοριακό, που δημιουργεί ενδεχομένως ακόμη περισσότερο ε, ακόμη περισσότερες περιπτώσεις ε, ε, κατάστασης μαζικής ζημίας που επίσης λαμβάνεται υπόψη αναμένουμε την αύξηση των αριθμών των διασυνοριακών τέτοιων περιπτώσεων ε, μαζικής ε, ζημίας. Η έκθεση ε, βασίστηκε στις πληροφορίες που ζητήσαμε να μας υποβάλουν τα κράτη-μέλη σε σχέση στις, στη δημόσια, το δημόσιο αίτημά μας για συλλογή πληροφοριών ε, και ε, στα δεδομένα ε, της μελέτης που συνοδεύει την αξιολόγηση. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τη μελέτη αυτή η οποία αναφέρεται και στην έκθεση. Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς ε, να ε, έχει πρόσβαση σε αυτήν ε, την μελέτη, αλλά ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες να είναι διαθέσιμη. Την περασμένη εβδομάδα με τον ανάδογο του έργου προσπαθήσαμε να χτενίσουμε την έκθεση αυτή προκειμένου να είναι διαθέσιμη, αλλά είναι πάνω από 1200, 1200 σελίδες. Ελπίζω πάντως ότι θα μπορείτε σύντομα να την προσπελάβνετε στην ιστοσελίδα τη γενική διεύθυνση Just. Να περάσω τώρα στα βασικά πορίσματα τη έκθεση που πιστεύω ότι αντανακλούν και τη, κάποια στοιχεία των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάποια στοιχεία δηλαδή έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή πριν από την έγκριση της σύσταση. Πρώτον, ένα από τα κύρια αναμενόμενα ζητήματα που είναι το, η νομοθετική παρακολούθηση ε, η οποία ήταν ε, περιορισμένη. Ε, είδαμε πολλά κρατημέλη μετά την έγκριση της σύστασης τα οποία προσάρμοσαν, τροποποίησαν ή εισήγαγαν τέτοιου είδους μηχανισμούς συλλογικής ενδικής προστασίας. Δεν λέω ότι η τροποποίηση αυτή είναι πάντοτε συμβατή με τις ε, αρχές της σύστασης. Ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η συλλογική ένδικη προστασία καλύπτει και τις δύο μορφές της προστασίας αυτής, δηλαδή έχουμε τα ασφαλιστικά μέτρα και έχουμε και τις αποζημιώσεις και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με τα ασφαλιστικά μέτρα υπάρχει, υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα η οδηγία περί ασφαλιστικών μέτρων που ισχύει στην περίπτωση ε, παραβίασης των δικαιωμάτων του καταναλωτή η οποία εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη με ικανοποιητικό μη τρόπο. Ε, οι συνάδελφοι που έκαναν την σχετική αξιολόγηση ξέρετε ότι προετοιμάζουν αυτήν την, τη, τη βελτίωση της ε, οδηγίας αυτής περί ασφαλιστικών μέτρων. Τα ασφαλιστικά μέτρα υπάρχουν λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, στον τομέα του καταναλωτικού δικαίου, Όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα ε, σε, σε, σε άλλους τομείς, δεν υπάρχει τέτοια ομοιογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ε, της, ε, των ασφαλιστικών μέτρων σε άλλους τομείς πέραν του καταναλωτικού δικαίου. Ε, όσον αφορά τώρα την, το ευαίσθητο θέμα της αποζημίωσης, ε, υπάρχει σε 19 κράτη-μέλη, που σημαίνει ότι σε 9 κράτη-μέλη δεν είναι δυνατό για τους ε, ε, ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις μαζικής ζημίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υποφεληθούν από την συλλογική αποζημίωση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, εντάχει, γιατί πιστεύω ότι η έκθεση ε, είναι εύκολο να ε, διαβαστεί. Είναι μόνο 22 σελίδες και έχει, περιλαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες. Απλώς θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποια σημεία. Κάτι το οποίο αναγνωρίζεται ως βασικό σε σχέση με την ε, καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση αυτής είναι το να ε, εξασφαλίζεται το παραδεκτό της αγωγής κάθε φορά. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται να είναι πολύ προβληματικό στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, όλοι όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους μηχανισμούς ε, έχουν κάποιους μηχανισμούς που επιτρέπουν την απόρριψη μη παραδεκτών αγωγών. Uh, Ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα είναι αυτό της ε, συλλογικής αγωγής και της διαφορετικής μορφής που μπορεί να λάβει. Μία από τις πιο ε, βασικές μορφές είναι η αντιπροσωπευτική. Δηλαδή κάποιος εκπροσωπεί όλους όσους ε, έχουν πληγεί από αυτήν τη μαζική ζημία... Ε, Υπάρχει λοιπόν ένας φορέας που εκπροσωπεί τους ανθρώπους αυτούς, όμως πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Το κράτος μέλος ε, που προβλέπει τέτοιου είδους ε, διαδικασία θέτει κάποιους ε, όρους και προϋποθέσεις που πάλι ποικίλουν σε, μεταξύ των κρατών μελών από πολύ ε, αυστηρές μέχρι πολύ λιγότερο αυστηρές Κάτι το οποίο ενδεχομένω να δημιουργεί τον κίνδυνο ότι αυτές, αυτοί οι φορείς εκπροσώπησης ε, ε, δεν ε, είναι έγκυρη, έγκυρος φορέας γιατί δεν πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις αυτής της ε, διαδικασίας που προβλέπει το κράτος μέλος. Υπάρχει επίσης και το opt-in και το opt-out. Η επιλογή συμμετοχής ή μη. Υπάρχει ο μηχανισμός αναγνώρισης των μελών της ομάδας. από τα κράτη-μέλη που προβλέπουν ε, την αποζημίωση, κάποια κράτη-μέλη αποκλειστικά εφαρμόζουν συμμετοχή Καταρχήν, δηλαδή ότι κάποιος πρέπει να δηλώσει ότι θέλει να συμμετέχει σε μια συλλογική αγωγή αν έχει υποστεί μαζική ζημία ε, και για όσους, ε, για όσους ισχύει και το opt-in και το opt-out Πρέπει να δηλώσει κανείς ότι ε, θέλει να ακολουθήσει το opt-out. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί μάλλον περισσότερο με τη διαδικασία ε, opt-in, έχουμε δει και περίπτωση καταχρηστικής προσφυγής ε, στη δικαιοσύνη και στην περίπτωση opt-out. όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την αρχή της κάλυψης ε, των εξόδων ε, από το μέρος που θα χάσει τη δίκη, βάσει της αρχής ότι αυτός που χάνει πληρώνει, ο χαμένος πληρώνει. όμως, ε, οι λεπτομέρειες, οι τρόποι εφαρμογής είναι αυτές που συνθέτουν το βάρος που, έχει να, που πρέπει να φέρει το μέρος που χάνει τη δίκη και που αυτό διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Δηλαδή τι θα πει ακριβώς αποζημίωση σε μία ε, αστική ε, αγωγή που επίσης διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ένα άλλο επίμαχο ζήτημα που το καλύπτουν οι συστάσεις και βεβαίως και η έκθεση είναι η χρηματοδότηση από τρίτο μέρος και τα έξοδα δικηγόρου, η αμοιβή του δικηγόρου. Αυτό αφορά κυρίως τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν, δηλαδή πολύ χαλαρές προϋποθέσεις οι οποίες σκοπό έχουν κυρίως να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια να είναι σαφές δηλαδή από πού προέρχεται η χρηματοδότηση, ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του χρηματοδότη και των μερών. Αυτό είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο στην Ευρώπη και είναι κάτι που δεν καλύπτει η νομοθεσία των κρατών μελών καθόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, συνέχιση της σύστασης αυτής ε, και εφαρμογή της πουθενά, ε, γιατί είναι ένα εντελώς καινούριο φαινόμενο. Το θέμα των εξόδων δικηγόρου έχει να κάνει με αυτό το θέμα της χρηματοδότησης ε, τρίτου μέρους, ε, γιατί τα έξοδα των δικηγόρων είναι ένα σημαντικό τμήμα του κόστους ε, της συλλογικής αγωγής. Επιτρέπεται σε νέα κράτη-μέλη, αλλά πηγαίνουν από 15% σε 50% για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα άλλα 18 κρατημέλη έχουν αυτό το σύστημα εξόδων, δηλαδή κάλυψη των εξόδων των δικηγόρων, η οποία εξαρτάται από το αποτέλεσμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Σημειώσαμε ότι 19 κρατημέλη έχουν ε, μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών συλλογικές, κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Υπάρχουν όμως κάποιες ιδιαιτερότητες. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι πολλές συλλογικές αγωγές επιλύονται χωρίς ε, προσφυγή σε κανέναν εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών. Το ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος μου, οπότε θα πάω ευθύ αμέσως στα συμπεράσματα. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης πρακτικής εφαρμογής των συστάσεων είναι, ε, αποκρισταλώνεται σε τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η σύσταση εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή της ε, περαιτέρω. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και θα υπάρξει ένα λεπτομερέστερο σχέδιο δράσης σχέση με το τι θα κάνουμε στο μέλλον με τις αρχές της σύστασης. Ειδική, ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στη χρηματοδότηση τρίτου μέρους. Ε, θέλουμε να μάθουμε λίγο περισσότερο, περισσότερα για το θέμα αυτό και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και τρίτο, συμπεράσματα, τρίτο συμπέρασμα, το προφανές πόρισμα ότι οι περισσότερες καταστάσεις μαζικής ζημίας στην Ευρώπη αφορούν τους καταναλωτές. προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξασφαλίζεται σε αυτή την περίπτωση μαζική ζημία, πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική παρακολούθηση. Αυτό τώρα είναι ε, σε στάδιο προετοιμασίας. Ο πρόεδρος Γιούγκερ το είχε αναφέρει ως τμήμα του New Deal για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Στέφαν Βόιτ, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λέβεν και θα μας μιλήσει για τη σύσταση του 2013. Έχετε 15 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση εντάχει θα ήθελα να πω ότι είμαι ακαδημαϊκός και θα κάνω ένα βήμα πίσω και θα σας μιλήσω για την ευρύτερη εικόνα. Ε, είχα ασχοληθεί με την συλλογική αγωγή του 14 από τους καταναλωτές μετά από μαζικές καταστροφές, για μαζικές καταστροφές και τα τελευταία χρόνια μαζεύω στοιχεία για τις συλλογικές ευρωπαϊκές αγωγές και κοιτάξαμε και άλλες τεχνικές συλλογικής προσφυγής ένδικα μέσα. Θα σας μιλήσω γενικά, θα κάνω πέντε παρατηρήσεις που ε, ίσως θα εμπνεύσουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη συλλογική προσφυγή σε ένδικα μέσα. Είναι ένα διφορούμενο ζήτημα, επηρεάζουν τα λόμπι και φαίνεται ότι το διακύβευμα είναι υψηλό. Αν δείτε τι συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση για τα συλλογικά ένδικα μέσα εγκλωβίζεται σε αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή πρόκειται για πολιτικούς συμβιβασμούς για να συμφιλιώσουμε αντιδίκους, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο που δεν είναι και ο πρωταρχικός στόχος Πολλές φορές θεωρούμε ότι ο ίδιος κίνδυνος ελοχεύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά την σύσταση του 13, πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για πολιτικό συμβιβασμό που βασίζεται στη ρεαλιστική κρίση ότι τίποτα άλλο δεν είναι δυνατό. Πρόκειται για ένα ποτ που ε, αντιφατικών στοιχείων που δεν θα μπορούσαν να συγκλίνουν διαφορετικά. Πολλές φορές εμείς οι ακαδημαϊκοί μπορούμε να είμαστε και αφελείς. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους. Ένας στόχος που αποκλείεται εξ αρχής, και αυτό είναι θετικό, είναι να αποφύγουμε τις συλλογικές ε, αγωγές ως μηχανισμούς πίεσης. Μετά θα πρέπει να δούμε ευρύτερα από τη μελέτη αντικτύπου του Οκτωβρίου του 2017 είναι, έχει πολύ συσταλτική ερμηνεία και γι' αυτό θα φτάσουμε σε συμπεράσματα τα οποία δεν είναι κοσμογονικά, αλλά έχουν σημασία. Η δεύτερη επιλογή είναι η αδράνεια. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η σύσταση έχει επικριθεί, αλλά πιστεύω, όπως είπε ο κύριος Γκάσκα, ότι ήταν ένα πολύ καλό ε, πνευματικό εγχείρημα διότι ορίζει αρχές και δικλείδες ασφαλείας και για εξοδικαστικές επιλύσεις μαζικών καταστροφών. Και όπως είπε και ο κύριος Γκάρσκα, οι περισσότερες αρχές δεν τηρούνται από τα κράτη-μέλη. Γιατί? Αυτό έχει να κάνει με, με το νομικό πολιτισμικό υπόβαθρο των 28 κρατών μελών. Κάτι που επηρεάζει τα επιμέρους στοιχεία καθώς ε, και την ευρωστία και την αδυναμία των συλλογικών αυτών μηχανισμών. Οι Ολλανδοί <coughs> θέλουν εξοδικαστική επίλυση οι Βέλγοι και Γάλλοι λαμβάνουν ε, υπόψη τις συλλογικέ αγωγές, ενώ στη Σκανδιναβία ο δημόσιος τομέας παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση διαφορών και φυσικά ε, είναι ουτοπικό να θέλουμε να συγκλίνουν όλα αυτά. Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν συλλογικό μηχανισμό χρήσης ένδικων μέσων και υπάρχει μια τέτοια πρόταση της Επιτροπής για ασφαλιστικά μέτρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά δομικά στοιχεία. Με βάση την εμπειρία μου, όλα ευσταθούν ή, ή, ή όχι από δύο δομικά στοιχεία. Το θέμα, το πρώτο θέμα είναι το μόνιμο θέμα. Δηλαδή ποιον εμπιστεύεστε να υποβάλει, να προσφύγει στη δικαιοσύνη τη στιγμή που η απόφαση θα τον επηρεάσει άμεσα. Σε περίπτωση αποζημίωσης, ποιος είναι, ποιος είναι ο μοχλός που θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιήσει το δικαστικό σώμα. Υπάρχουν ε, ad hoc οντότητες που θα μπορούσαν να δράσουν. Υπάρχει ανταγωνισμός. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που σχετίζονται με την πεντουσία οποιοδήποτε συλλαγικού μηχανισμού ενδικών μέσων. Το θέμα της χρηματοδότησης που σχετίζεται άμεσα με το προηγούμενο είναι πιο σημαντικό. Αν δείτε τον ε, μηχανισμό συλλογικών ενδίκων ε, μέσων στα κράτη-μέλη και αν μιλήσετε με επιχειρήσεις ενός καταναλωτών ή ε, δικηγόρων, βλέπετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση αυτών των μηχανισμών και τα κράτη-μέλη δεν έχουν κανόνες. Στο Βέλγιο θεωρήσαμε αφελώς ότι θα ισχύσουν οι κανόνες που ισχύουν σε ε, μία προσφυγή. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Επίσης ε, έγινε λόγος για χρηματοδότηση μέσω ενός τρίτου αντιδίκου. Όλες όμως οι συλλογικές αρρωγές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από έναν τρίτο αντιδικό όπως ισχύει στην Αυστραλία. Και φαίνεται ότι θα υπάρχει περισσότερη έρευνα αυτού του ζητήματος γιατί ίσως γίνονται και καταχρήσεις. Προσωπικά αν ε, δω αυτή την περίπτωση χρηματοδότηση από τρίτους, δεν υπάρχουν καταχρήσεις γιατί οι μηχανισμοί φιλτραρίσματος είναι πολύ καλοί. Οι επιχειρήσεις ε, δεν θα χρηματοδοτήσουν ε, ανούσιες αρρωγές, ανούσιες διαφορές, αλλά δεν χρηματοδοτούν αγωγές καταναλωτών γιατί δεν έχουν να βγάλουν πολλά χρήματα από αυτό. Άρα ε, ασχολούνται με το καθαρά επενδυτικό σκέλος. Το άλλο, το τέταρτο στοιχείο που ίσως είναι αντιφατικό, αλλά εμείς οι ακαδημαϊκοί είμαστε αντιφατικοί, οδηγεί στο εξής ε, συμπέρασμα. Έχω ασχοληθεί με συλλογικές αγωγές, αλλά υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί στα κράτη-μέλη για τη συλλογική προσφυγή σε ένδικα μέσα. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια υπέρ των καταναλωτών από τον συνήγορο του πολίτη, που προωθούνται από το συνήγορο του πολίτη. Επίσης υπάρχει η ρυθμιστική χρήση ένδικων μέσων και αυτό γίνεται από τις ε, ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπως στην περίπτωση της Σκανδιναβίας, Βελγίου, Ιταλίας και Ολλανδίας. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να γίνει χρήση συλλογικών ένδικων μέσων με χαμηλό κόστος. Δηλαδή μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ε, συλλογικές διαφορές για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές που επιλύονται μέσα στα πλαίσια μίας διαφοράς. Και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, δεν λέω ότι αυτό είναι το ε, Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά στην όλη συζήτηση της ε, συλλογικής χρήσης ένδικων μέσων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις συνιστώσεις όταν ορίζουμε την πολιτική μας, γιατί είναι εύληπτες και λειτουργικές πολιτικές. Εάν μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέμε πολλές φορές αυτή είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου ή άλλης Επιτροπής ή άλλης Γενικής Διεύθυνσης. Τέλος, αυτές οι τεχνικές είναι αντιφατικές. Έχουν υπέρμαχους και αντίμαχους και στο θέμα της ρυθμιστικής χρήσης ενδίκων μέσων χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και μηχανισμοί αναθεώρησης. Οι τεχνικές αυτές δεν ήταν απόρρια μια στοχοθετημένης πολιτικής αναπτύχθηκαν από τους τομείς καθεαυτούς. Γιατί πολλές φορές ο δικαιοδοτικός τομέας δεν λειτουργεί. Δηλαδή ε, κινούνται από τους ίδιους τους μηχανισμούς της αγοράς. Τέλος, η πέμπτη που παρατήρηση, και εδώ μιλάμε για μία ιδεώδη κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε μία, ένα ολιστικό πλαίσιο επίλυσης διαφορών με βάση τη χρήση συλλογικών ενδικών μέσων, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε όλα, όλες τις επιλογές για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών. Δεν μιλάμε για ε, ε, διαφορά του άσπρου από το μαύρο, ψωμί, το, το μαύρο ψωμί, αλλά το πώς θα ζυμώσουμε αυτό το ψωμί, πώς θα το παρασκευάσουμε. Αυτή Αυτά είναι μικρά αλλά ρεαλιστικά βήματα. Ορισμένα παραδείγματα υπάρχουν, δηλαδή οι συλλογικές ε, αγωγές έναντι του δημοσίου τομέα. Στην Φιλανδία μίλησα με τον εθνικό ρυθμιστή ή συνήργορο και μου είπε ότι χρησιμοποιεί αυτό το μηχανισμό μέσα στα πλαίσια της ε, ευρείας εργαλειοθήκης του. Το δεύτερο παράδειγμα ε, επιτρέπει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα εξοδικαστικά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε ασφαλιστικά μέτρα για να λάβουμε υπόψη και τις αστικές αγωγές, έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να μπορέσουν να αντιδράσουν μέσα στα πλαίσια της αρχής των εναλλακτικών, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ε, άλμα για τους ε, καταναλωτές. Και υπολείπεται 1,5 λεπτό από την παρουσίασή μου που σας χαρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Και περνάμε στο τρίτο μέρος της ακρόασης ποια είναι η άποψη των ενδιαφερομένων αφαιρών. Κυρία Αγκούστα Μάλκεβιτσιούτη, που είναι ανώτατη νομική σύμβουλος ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών, να λάβει το λόγο. Να σχολιάσει την έκθεση της Κομισιόν και να μας μιλήσει για τα επόμενα βήματα. Έχετε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας προσκάλεσε στην σημερινή συζήτηση. Πρέπει να πω ότι και η Επιτροπή σας αλλά και το δικό μας γραφείο τα τελευταία 30 χρόνια εργαζόμαστε πάνω στο θέμα της συλλογικής ένδικης προστασίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς και προτεραιότητα για τις οργανώσεις μέλη της BUC. Λυπούμεθα που εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό για την πρόσβαση των Ευρωπαίων καταναλωτών ε, στη δικαιοσύνη. Πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Γκάρτσκα, ε, υπάρχει ένα, μια εμβαλωματική ε, εικόνα σε ό,τι αφορά τις εθνικές αντισταθμιστικές διαδικασίες ένδειξης προστασίας. Λίγες διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά. Τα κενά των δυνατοτήτων ένδικης προστασίας στην Ευρώπη τα είδαμε ξεκάθαρα στην περίπτωση της ε, υπόθεσης Volkswagen που τη γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες υποθέσεις ε, σε κράτη-μέλη αλλά και διασυνορικές όπου οι καταναλωτές μένουν με χέρια ενώ εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες ε, ευρώ είναι η συνολική ζημία πέραν της απογοήτευσης και της αδικίας που νιώθουν οι καταναλωτές, ε, το αποτέλεσμα ε, του χάσματος του κενού αυτού είναι ότι είναι πολύ λίγος και ο πολύ μικρός αποτρεπτικός ε, χαρακτήρας και δεν αποτρέπονται αυτές οι πράξεις, δηλαδή παραβίαση των καταναλωτικών δικαιωμάτων. Χρειάζεται λοιπόν, όπως φαίνεται και από την εμπειρία μας, μια ειδική διαδικασία για ένδικη προστασία, συλλογική. δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την αλλακτική επίλυση διαφορών. Γιατί είδαμε ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν κίνητρα να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εναλλακτικό μηχανισμό ή να ξεκινήσουν ε, ε, τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού. Και από τις ε, βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, που εν γέννη λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα αλλακτική επίλυσης διαφορών, αλλά έχουν και διαδικασίες Συλλογική ένδικης προστασίας, είναι και αυτό μια δυνατότητα που προβλέπεται στο δίκαιό τους. Η επιβολή από, την, από το κράτος, ούτε και αυτό λειτουργεί πάντοτε, γιατί πολλές φορές είναι λίγες οι αρμοδιότητες και δεν μπορούν να επιβάλλουν στον εμπόρο να πληρώσει. Έγινε μια προσπάθεια εθνικές καταναλωτικές αρχές να έχουν αυτή τη ε, δυνατότητα να εξασφαλίζουν την ε, αποζημίωση ή τέλος πάντων να ζητούν από τον έμπορο να καταβάλει αποζημίωση. Αλλά τα κράτη-μέλη ήταν ε, αντίθετα. Γι' αυτό και η πρόταση σχετική απαλήφθηκε από την πρόταση του Συμβουλίου τελικά της Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα άλλα ένδικα μέσα. Ξέρετε επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σαφή πλειοψηφία μεταξύ των πολιτικών ομάδων ζήτησε να υπάρξει ένας μηχανισμός συλλογικής ένδικης προστασίας πέρυσι τον Απρίλιο στο ψήφισμά του για τι μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητομηχανίας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα να έχουμε δεσμευτική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε τα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν να θεσπίσουν συλλογικές διαδικασίες αποζημίωσης. Έχουμε παραδείγματα από κάποια κράτη-μέλη όπως το Βέλγιο, την Ιταλία ή την Πορτογαλία. Εκεί πράγματι υπάρχουν λειτουργικά αποτελεσματικά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό με την αναθεώρηση της οδηγίας περιασφαλιστικών μέτρων. Δεν θα είναι βέβαια ακριβώς ε, ένας μηχανισμός συλλογική ένδειξης προστασίας, αλλά είναι μια επιλογή την οποία υποστηρίζουμε, διότι θα βελτιώσει ήδη σημαντικά την κατάσταση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, που είναι θύματα αθέμητων πρακτικών. Επίσης, ε, αν έχουμε καταλάβει καλά την πρόθεση της Κομισιόν, αυτή η απόφαση για την αποζημίωση θα γίνει μετά την ε, επιβολή ασφαλιστικών μέτρων όταν έχει αποδειχθεί ότι παρεύει τον νόμο ο έμπορος. Και στην περίπτωση αυτή είναι λογικό να υπάρξει αποκατάσταση στην προτέρα της ε, παράβασης αυτής κατάσταση. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ε, να μην ισχύουν κάποιες ρήτρε, οπότε θα πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές. Γι' αυτό ή θα πρέπει τα ποσά τα οποία σπράχθηκαν παρνόμως να τους επιστραφούν. Έχουμε περιπτώσεις Τέτοια αποκατάστασης στις παραδόσεις των κρατών μελών, στι νομικέ παραδόσεις. Τι ζητούμε τώρα με αυτό το εργαλείο. Σε ό,τι αφορά, το πεδίο των διαδικασιών συλλογικής ένδειξης προστασίας, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς ενδιαφέροντος για τους καταναλωτές, όπως είναι ο ανταγωνισμός και η υγεία. Διότι υπήρξαν υποθέσεις στην Ευρώπη που υπήρξε ζημία λόγω κάποιου φαρμάκου, βλάβη ή κάποιας, ε, κάποιο το τεχνολογικό προϊόντος. Οι καταναλωτές όμως δεν κατάφεραν να πάρουν αποζημίωση. Οι ενώσει των καταναλωτών πρέπει να είναι μεταξύ των φορέων που θα είναι σε θέση να δρομολογούν διαδικασίες ε, τέτοιων προσφυγών και σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο και θα πρέπει να υπάρχει ελάφρυνση του κόστου. δηλαδή να τροποποιηθεί η αρχή του οδηγητής διάδικο πληρώνει, για να μπορούν οι ενός καταναλωτών να αναλάβουν δράση. Αυτό ήδη είναι εφικτό σε Πορτογαλία, Μάλτα, Ισπανία και Ιταλία και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν από αυτό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, το είπε και ο καθηγητής Βουτ, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ευρείες δυνατότητες χρηματοδότησης. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, κρατικής χρηματοδότησης, ε, κάποιων τελών ε, συμμετοχής, δωρεές, χρηματοδότηση έργου, δραστηριότητες πώληση ή συμβουλευτικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση από τρίτων και αυτό το τελευταίο πρόσφατα Ορισμένοι αμπικομένοι, το χρησιμοποίησαν ως ένα παράδειγμα για να καταδείξουν τους κίνδυνους και τις πιθανές καταχρήσεις των διαδικασιών συλλογικής ένδικης προστασίας. Ωστόσο, η εμπειρία των μελών μας ε, είναι αντίθετη με τους ισχυρισμού αυτούς. Για παράδειγμα, το αυστριακό μέλος ε, της οργάνωσής μας χρησιμοποιεί αυτή τη χρηματοδότηση ήδη από το 1994 και τους βοήθησε να εξασφαλίσουν εκατομμύρια ευρώ αποζημίωσης για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, μεταξύ των ετών 2011 και 2014, το αυστριακό μέλος ε, της ε, οργάνωσής μας εξασφάλισε 55 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για τους καταναλωτές χρησιμοποιώντας τις συλλογικές προσφυγές αυστριακού τύπου. Βέβαια, η καθού ε, θέλουν μια προμήθεια για τον ε, κίνδυνο, για το ρίσκο που αναλαμβάνω, πολλές φορές ε, όταν υπάρχει ένας δεκανονισμός συμφωνούν να πληρώσουν ε, το τέλος και επομένως παίρνουν την πλήρη αποζημίωσή τους οι καταναλωτές. Επίσης, πολλές φορές οι χρηματοδότες αυτοί δίνουν πολύτιμη νομική ε, πληροφόρηση μέσω της εμπειρίας που έχουν στο δίκαιο της αλλοδαπής, επαφές τους για τη μετάφραση κτλ. Επίσης πολλές φορές ε, προσφέρουν και περαιτέρω χρηματοδότηση κάτι σημαντικό για τις ενώσεις καταναλωτών που δεν έχουν τόσο μεγάλη χρηματοδότηση. Σίγουρα πολλές φορές οι διαδικασίες οι δικαστικές ε, γίνονται μακροχρόνιες, ε, δεν είναι επιτυχής πολλές φορές η έκβασή τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε να αναπτύξουμε αυτούς τους μηχανισμούς ασύλλογης ένδειξη προστασίας, γιατί είναι λογικό, καθότι πρόκειται για κάτι καινούριο. Χρειάζεται νομοθεσία και εμπειρία και για τους δικηγόρου, για τους δικαστές ε, και για τους διαδίκους να συνηθίσουν τις νέες διαδικασίες και να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. και μόνο όταν υπάρχουν ε, αυτές οι δικαστικές διαδικασίες θα, μπορούν ε, να, ε, θα μπορεί να αξιοποιηθεί και το πλήρες δυναμικό των φιλικών διακανονισμών ή της αποζημίωσης μέσω αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω τώρα τον κύριο Πέδρο Ολιβέηρα να πάρει το λόγο. Από την Business Europe, Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων. Θα μας πει και ο κύριος τα σχολεία του. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί καλέσατε τη Business Europe. Η Business Europe είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός ομπρέλας με μέλη από 33, 33 κράτη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμαστε εδώ και 30 χρόνια ε, όπως οι συνάδελφοι από την ΜΠΕΟΚ για τη, με τις συλλογικές αγωγές, μας ενδιαφέρει βεβαίως να, να εφαρμοστεί καλύτερα το δίκαιο των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις ε, δρούν διαχρονικά. Γι' αυτό είναι προς συμφέρον τους να δικαιώνονται οι καταναλωτές τη στιγμή που τα αγαθά δεν συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές. Ε, θα γνωρίζετε βέβαια ότι είμαστε μία από εκείνες τις φωνές που τάχθηκε κατά ενός συστήματος συλλογικών προσφυγών σε ένδικα μέσα. Υπάρχουν θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας, περιορισμού των συνθήκων και δεν υπάρχουν στοιχεία για μια ευρύτερη εμβέλεια υποθέσεων ή διαφορών που το επιβάλλουν. Θεωρώ ότι ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες έχουν τεθεί ήδη από το 2012 γι' αυτό για μας. Δεν είναι θέμα η αποζημίωση, αλλά πώς μπορεί να παρασχεθεί αποτελεσματικότερα. Και οι υποθέσεις, μάλλον τα συστήματα της Πορτογαλίας και της Ιταλίας δεν είναι αποτελεσματικά. Εγώ πιστεύω το αντίθετο, γιατί αν δείτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τη δράση του, βλέπετε ότι χρειάζεται μία διετία για επίλυση διαφοράς. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Ήμουν ε, δικηγόρος στην ε, Πορτογαλία και το ξέρω από πρώτο χέρι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ε, η συνειδητοποίηση και η χρήση των μέσων που είναι πιο αποδοτικά και λιγότερο δαπανηρά. Γι' αυτό δεχτήκαμε και την εναλλακτική επίλυση διαφορών, επίλυση των μικροδιαφορών και την ε, οδηγία περί εντολών για ασφαλιστικά μέτρα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν ε, μέτρα για ε, συλλογική χρήση των ένδικων μέσων, γιατί τη συλλογική, ένδειξη, ένδικη συγγνώμη, προστασία στους προσεχείς μήνες. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι τα συμφραζόμενα λοιπόν δράσεις και κάτι που ανέφερε ο κύριος Βουτ που είναι η εφαρμογή στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Και τέλος θα μιλήσω για τις δικλίδες ασφαλείας που είναι επιτακτής και ανάγκης σε μας τον επιχειρηματικό κόσμο. Πώς ε, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με, με τους μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας, ακόμα από αμερικανικές εταιρείε, το τι ακριβώς συμβαίνει και σπάνια οι συλλογικές αγωγές φτάνουν σε αυτά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Επίσης, από το Γραφείο Χρηματοοικονομικής Προστασίας στην Αμερική βλέπουμε ότι ο καταναλωτής παίρνει μία αποζημίωση, μέση αποζημίωση 32 δολαρίων, ενώ ο συνήγορος ένα εκατομμύριο δολάρια. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Πολλές φορές οι καταναλωτές κατά 85% δεν λαμβάνουν καν αποζημίωση και πολύ συχνά, ακόμα και να λάβουν αποζημίωση, η αξία είναι χαμηλότερο από το ίδιο το γραμματόσημο. Αλλά αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Ε, στις ΙΠΑ το βλέπουμε και στην ε, Αυστραλία όπου οι καταναλωτές λαμβάνουν αποζημίωση μερικά λεπτά του δολαρίου. Και αυτό το θέμα λοιπόν η ε, και η κινητήριος, δύναμη στην επίλυση διαφορών στις ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κατάχρηση αυτής της επίλυσης διαφορών, αλλά η σύσταση δεν αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις που συνδυαστικά μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι παράλληλο με αυτό. Τον είπα, η χρηματοδότηση αυξάνεται και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 23 τέτοιες περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και 16 στην Ολλανδία. Η Ολλανδία υπάρχουν 17 ε, δις προς επένδυση και πασχίζουν να δουν πού θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτές οι δύο χώρες, γιατί σε αυτές τις δύο χώρες, γιατί σε αυτές, αυτές οι δύο χώρες προσπαθούν να επιλύσουν διεθνείς διαφορές, κάτι το οποίο τις καθιστά δελεαστικές για αυτά τα επιχειρηματικά πρότυπα και μοντέλα. Γιατί ε, επιτρέπουν ένα 100 με 250% ε, αποζημίωση και απόδοση. Μιλάμε λοιπόν για συλλογικούς ε, ένδικους μηχανισμούς όπου ε, έχουμε ε, να κάνουμε μεσορία καταναλωτών και υπάρχει opt-out, διαδικασία opt-in και opt-out όσον αφορά εταιρείε συνηγόρων και ούτω καθεξής. Και όπως είπε και η Επιτροπή, 19 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς συλλογικής ενδικής ε, προστασίας. Αλλά υπάρχει επιλεκτική χρήση των ε, δικλείδων ασφαλείας και βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν γίνεται σωστή χρήση των δικλείδων ασφαλείας. Το δεύτερο σημείο που αφορά την εφαρμογή από τον ε, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισονομία και ο κυρωτικός μηχανισμός θα πρέπει να αποτελέσει προνόμιο του δημοσίου τομέα. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως στη Γερμανία όπου η πλειοψηφία ε, αφορά ε, εφαρμογή από τον δημόσιο τομέα. Άρα πολλές φορές υπάρχει ολίσθηση ε, εφαρμογής. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις αποτυχίες της αγοράς. Τρίτο και τελευταίο σημείο αφορά τις δικλείδες ασφαλείας είναι επιτακτικές και στην ε, μελλοντική πρόταση περιμένουμε ένα αυστηρό πλαίσιο δικλείδων ασφαλείας κατά των καταχρηστικών διαφορών. Ήδη υπάρχει ένας ελάχιστος ε, παρονομαστής στη σύσταση του 2013, άρα δεν θα ε, δράσουμε προς τα πίσω, δεν θα παλινοδίσουμε. Μέσα σε δύο λεπτά θα ήθελα να μιλήσω για το ότι ε, αυτός που χάνει πληρώνει. Είμαστε υπέρ του opt-in επίσης, της ε, πιστοποίησης, γιατί στην Πολωνία η διαδικασία πιστοποίησης ήταν πολύ αυστηρή, αλλά τώρα ε, έχει αποδυναμωθεί Επίσης, τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να περιοριστούν και θεωρούμε ότι, να, ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει το forum shopping, γιατί για τις Βρυξέλλες ένας κανονισμός δεν αρκεί. Εάν εμπίπτει σε μία συγκεκριμένη δικαιοδοσία, θα πρέπει να ξέρουμε πώς εξελίσσεται και ε, ο καθηγητής Βουτ μίλησε για κάτι πολύ σημαντικό, για το ποιος μπορεί να προωθήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ζωτικής ε, σημασίας για μας. Μιλάμε για ε, οντότητες ε, που έχουν που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Πρόκειται για οργανισμούς που δρούν στα κράτη-μέλη, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους τους φορείς που προβάλλουν ε, αξιώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ αυστηροί εδώ σε σχέση με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τη διαφάνεια, καθώς και άλλα στοιχεία. Τέλος, ε, χρηματοδότηση από τρίτους, ως προς αυτήν αποτελεί μεγάλη ανησυχία. Η Μπόκ λέει ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία πολλές φορές, αλλά πρωταρχικός στόχος είναι η απόδειση της επένδυσης. Δεν τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση των καταναλωτών. Αυτό θα μπορούσε να έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα και υπάρχουν ε, ρήτρες, συμβατικές ε, ρήτρες, που τους δίνουν ε, προνόμια μπορούν να εγκρίνουν ε, προσχέδια των διαδίκων και μπορούν να αμφισβητήσουν και την τελική απόφαση, την επίλυση της διαφοράς δηλαδή. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχουμε υψηλές προσδοκίες. Η Business Europe δεν ξέρει κατά πόσο χρειάζεται ένας τέτοιος συλλογικός μηχανισμός, αλλά θα συνεργαστούμε από πλευράς ε, επιχειρήσεων ως προς τους ε, καταναλωτές, έτσι ώστε να υπάρχουν αναλογικές λύσεις στα προβλήματα που εγκύπτουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στη συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ε, κύριε Ρέντα, Κυρία Ρέντα είναι πρώτη. Ε, παρακαλώ να είστε σύντομοι για να υπάρχει χρόνος για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ενδεχομένω και οι άλλοι προσκεκλημένοι να θέλουν να πάρουν το λόγο. Το νομικό μέσο που επιλέξετε. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε την αναθεώρηση της οδηγίας περί ασφαλιστικών μέτρων αντί για κάτι άλλο, γιατί εμείς δεν θέλουμε μόνο καταναλωτικό δίκαιο να καλύπτεται, ούτε μόνο τα αντισταθμιστικά μέτρα, αλλά και η αποζημίωση και άλλοι τομείς δικαίου. Θα είναι λοιπόν ενδιαφέρον να μας το πείτε αυτό και κάτι ακόμη, σε ποιο βαθμό η πρόταση αυτή θα είναι οριζόντια. Και δεν εννοώ με αυτό μόνο τους τομείς δικαίου που θα καλύπτονται, αλλά κατά πόσο το σχέδιο είναι να είναι ειδικό για ε, συγκεκριμένα νομοθετήματα ή αν θα είναι πραγματικά οριζόντιο, δηλαδή αν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε νομοθεσία. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι απαραίτητο, πολύ απαραίτητο να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί υπάρχουν ή ακόμη κάποια κράτη-μέλη που δεν έχουν κανένα σύστημα σχετικά, αλλά τι προσέγγιση θα έχουμε σε σχέση με την εναρμόνιση των κρατών μελών που ήδη έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Βέβαια, θέλαμε λοιπόν στο τέλος ε, της διαδικασίας ε, κάποια κράτη-μέλη να ε, αχάσουν διαδικασίες που είναι φιλικές προς το χρήστη. Ε, γιατί σε αυτή την περίπτωση το opt-out θα είναι χρήσιμο, γιατί αν σκεφτεί κανείς ε, τους κινδύνου για την υγεία από το Dieselgate, ε, ήταν μεγαλύτερη για τους ίδιου τους οδηγού. Και ακόμη και αν ε, κάποιος δεν το γνώριζε ότι το δικό του το ε, αυτοκίνητο ε, το δικό του το αυτοκίνητο το αφορά μια τέτοια συλλογική αγωγή μπορεί να επιλέξει να μην συμμετέχει. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα απαιτήσει όλοι να διατηρήσουν το opt-in ή θα επιτρέπει και το opt-out. Όσον αφορά το μετριασμό της κατάχρησης έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα ε, υποθέσεων της, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι καταχρηστικές όχι μόνο όπως γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, όχι επειδή υπάρχει μηχανισμός opt-out και καταναλωτικό δίκαιο δεν σημαίνει αυτό υποχρεωτικά ότι είναι μία κατάχρηση υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα κατάχρησης που θεωρείται ότι πρέπει να τα επιλύσουμε ή είναι ένας θεωρητικός φόβος για το μέλλον Ευχαριστώ κυρία Χάουτελα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω η εμπειρία από τις σκανδιναβικές χώρες, ειδικότερα από τη Φιλανδία, όπου η συλλογική αγωγή αφορά κυρίως καταναλωτικές υποθέσεις, έχει δηλαδή πολύ περιορισμένη εμβέλεια. Το ερώτημά μου λοιπόν έχει να κάνει και με αυτό που είπε η Γιούλια Ρέντα, κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο ε, σε αυτή τη φάση πριν μπούμε στην νομοθετική διαδικασία να συζητήσουμε την επέκταση σε άλλους σχετικούς τομείς. Δεν ξέρω ε, αν πρέπει οριζόντια να καλύψουμε τα πάντα, αλλά αναφέρομαι στην περιβαλλοντική υγεία, την ισότιμη μεταχείριση, τις ε, συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το ερώτημά μου, γιατί ε, Φοβούμαι ότι αν αρχίσουμε από ένα πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, ε, τότε θα είναι η, χρησιμότητα ε, της ένδικης προστασίας και πολύ περιορισμένη. Το ερώτημά μου αφορά επίσης και το φιλανδικό μοντέλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, που επισκεφτήκατε τον ε, φιλανδό συνήγορο του πολίτη, γιατί... Ε, έχει μια μεγάλη ευαισθησία σε σχέση με τα δικαιώματα ε, παρά το ότι το σύστημά μας αφορά περισσότερο το καταναλωτικό δίκαιο ε, όταν συμμετέχουν σε μια συλλογική αγωγή οι πολίτες μας δεν πληρώνουν εκείνοι η εταιρεία χάνει ή ο δημόσιος ε, τομέας χάνει. Ε, θεωρείτε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μεταφερθεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά συνεπώς τα κράτη-μέλη. Κάτι ακόμη σε σχέση με τη λογοδοσία των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τα θύματα ζημίας ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά τις ε, δραστηριότητες τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάω για παράδειγμα για μια δασοκομική επιχείρηση στην Γουατεμάλα ε, ή μια αγγλική εταιρεία που προκαλεί μια ζημία στα δικαιώματα αυτοχθόνων πληθυσμών ε, σε κάποια αφρικανική χώρα για παράδειγμα. Έχουμε βέβαια τις κατευθυντήρες γραμμές ε, του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εφαρμόσει τον τρίτο πυλώνα αυτών που είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα. Πιστεύετε μήπως ε, ότι παράλληλα με αυτό που συζητάμε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και αυτό το θέμα και να βρούμε έναν τρόπο να, να ε, εκπληρώσουμε και αυτή την υποχρέωσή μας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυμάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός ε, της Ένωσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως θα μπορούσαν οι εμπειρογνώμενες να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Κύριος Νόστερ πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. σα ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο πολύ διεξοδικές ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, την απάντησή μου ευχαριστώντας την Επιτροπή σας ε, γιατί πήρε την πρωτοβουλία της ε, συζήτησης αυτής και του διαλόγου αυτού σε σχέση τώρα με τα ερωτήματα που καλύπτουν προφανώς διάφορους τομείς. Θα αρχίσω καταρχάς με την έκθεση και μετά θα αφήσω τους συναδέλφους που ασχολούνται με την ε, νέα ε, πρωτοβουλία να συμπληρώσουν ε, τις λεπτομέρειες σε σχέση με την μελλοντική πρωτοβουλία. Το ερώτημα του πεδίου εφαρμογής της μελλοντικής πρωτοβουλίας και για ποιο λόγο, όπως αναφέρεται στην έκθεση, θα ήταν περιορισμένο μόνο στους καταναλωτές ή θα είναι τμήμα του New Deal για τους καταναλωτές. Συμπεράναμε στην έκθεση και στην ανάλυση μας ε, ότι οι περισσότερες περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν καλύπτουν την προστασία του καταναλωτή, συγκεκριμένα το θέμα των εκπομπών ε, ε, των αυτοκινήτων καλύπτουν κυρίως τους καταναλωτές και βάσει αυτών των πορισμάτων, κατά τη γνώμη μας, ε, ε, θα ήταν χρήσιμη μία ε, προσφυγή στο συγκεκριμένο τομέα. Σε σχέση τώρα βέβαια με το μέγεθος, ε, ε, με, την, με, την, ε, με το πεδίο εφαρμογή της, της διαδικασίας, θα αφήσω το συνάδελφο να πει περισσότερα, αλλά σε σχέση με το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση να προτείνει κάτι σε σχέση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη δικαιοδοσία των κρατών ε, και κατά πόσο επεκτείνεται σε επικόους τρίτων χωρών. Αυτό ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 και κατά, την, ε, κατά τις διαπραγματεύσεις αυτού του μέσου θεωρήθηκε καλό και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο να μην το καλύψουμε αυτό στον κανονισμό, αλλά πολυμερός σε ένα διεθνές φόρουμ. σε αυτή τη φάση μπορώ να σας πω ότι η διάσκεψη της Χάγης για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο έχει ένα ε, σχέδιο επέκτασης της δικαιοδοσίας των, της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων σε αυτή την περίπτωση, οπότε Αν δεν προχωρήσει αυτή, αυτό το εγχείρημα θα μπορούσαμε να καταφύγουμε όπως, αναφέρθηκε και, όπως αναφέρεται στο τέλος ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 1 και, ε, και να υπάρξει μια μονομερής δράση. Θα ήθελα τώρα οι συνάδελφοι να απαντήσουν ε, λεπτομερέστερα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστώ. Ιωάννα Πατράσκου και Αγγελίν Μπράουν, αν δεν κάνω λάθος, θα λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ. Για να συμπληρώσω αυτά που εξήγησε ήδη ο συνάδελφος, εμείς προβλέπουμε την αναθεώρηση της οδηγίας ε, περί ασφαλιστικών μέτρων ε, λόγω των πορισμάτων του ελέγχου καταλληλότητας ε, του καταναλωτικού δικαίου ε, ως προς την αποτελεσματικότητα του, ε, της ορισόντιας νομοθεσίας ε, περί καταναλωτών ε, και το κεκτημένο αυτής ε, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε βέβαια την αποτελεσματική εφαρμογή, δηλαδή να μπορούν οι καταναλωτές, καταναλωτές όντως να υποφεληθούν από τους κανόνες αυτούς. Ε, αυτή η τμήμα της προσπάθειας αυτής ε, είναι βέβαια να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της οδηγίας ε, ασφαλιστικών μέτρων που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς που πληρούν τις προδιαγραφές να εκπροσωπήσουν κάποιους ανθρώπους για να σταματήσουν την παραβίαση δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτές οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες όντως ε, σταματούν τις ε, παράτυπες δραστηριότητες των εμπόρων, ε, κάποιες έμεσες συνέπειες των πρακτικών αυτών παραμένουν και οι καταναλωτές εξακολουθούν να υφίστανται τη ζημία χωρίς να έχουν τη δυνατότητα μεμονωμένα να επιβάλλουν την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ένα λογικό επόμενο βήμα θα ήταν να διερευνήσουμε πώς και ε, αν θα έπρεπε να δούμε το θέμα της ε, ε, προστασίας στο πλαίσιο της οδηγίας περιασφαλιστικών μέτρων. Όπως ακούσαμε βέβαια σήμερα, είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα και υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη τις διαφορετικές νομικές ε, παραδόσεις των κρατών μελών βεβαίως, όπως επίσης και τα συμφέροντα όλων των μερών και των εμπόρων και των καταναλωτών. Συνεπώς, βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία ολοκλήρωσης αξιολόγησης αντικτύπου μας για να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω αυτό να σας δίνει κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το για ποιο λόγο αποφασίσαμε να καλύψουμε αυτό το θέμα στο πλαίσιο της οδηγίας περί μέτρων, όπως έχει αναθεωρηθεί αυτή στο πλαίσιο του New Deal για, τις, για τους καταναλωτές. Και κάτι ακόμη, για το πεδίο εφαρμογής και το κατά πόσο θα είναι περιορισμένο μόνο σε ζητήματα καταναλωτών, πράγματι αυτό είναι τμήμα των ε, στοιχείων που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, οι καταναλωτές και τα συμφέροντά τους καλύπτονται και την χάνουν προστασίας ε, όχι μόνο από την νομοθεσία κατά, την, περί, καταναλωτών, αλλά και από άλλα άλλες νομοθεσίες άλλων τομέων ε, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, οι τηλεπικοινωνίες ε, και σας αναφέρω τις πιο προφανείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για παράδειγμα. Το βλέπουμε λοιπόν και υπό αυτήν την οπτική γωνία για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή της ε, υφιστάμενης οδηγίας. Ευχαριστώ. Ε, Ο καθηγητής Φουτ. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα για το φιλανδικό μοντέλο. Ουσιαστικά είναι δύο. Τα μοντέλα ένα στη Φιλανδία που είναι όπως εσείς το περιγράψατε και είναι αρκετά στενό αν θέλετε, αλλά υπάρχει και το δανέζικο μοντέλο. Έχουμε έναν συνήγορο των καταναλωτών ο οποίος ε, είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει συλλογική προσφυγή opt-out. Αλλά Επαναλαμβάνω, είναι συνήγορος του πολίτη, συνήγορος του καταναλωτή. Δεν είναι παραδοσιακό συνήγορος του πολίτη, αλλά είναι μια αρχή επιβολή. Αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο με τα μοντέλα αυτά είναι πως οι φορείς αυτοί έχουν μια τεράστια εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία. Τελικά λοιπόν κάποιες φορές ε, με πιάνει η αλλεργία με αυτή τη συζήτηση περί κατά των ε, μηχανισμών ένδικης προστασίας. Φυσικά και χρειάζονται, απλά πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Λείπει όμως η συζήτηση για το ευρύτερο αυτό πλαίσιο. Αυτό που είναι λοιπόν πολύ θετικό στη Δανία για παράδειγμα είναι ότι ο τέος συνήγος του πολίτη που τώρα είναι γενικός αγγελέας υπό την πυρηνική βόμβα συνιστά ε, η μαζική προσφυγή opt-out. Είπε λοιπόν στην εταιρεία, φτιάξτε το τώρα, εγώ θα το ελέγξω, αλλιώς θα ρίξω την πυρηνική μου βόμβα. Και λειτουργήσε. Αν δείτε μελέτες περιπτώσεων που έχουμε συλλέξει, δουλεύει το σύστημα. Και σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι σκέφτεται ο κόσμος σε κουτάκια. Πρέπει να δούμε τη συνολικότερη εικόνα και να αξιολογήσουμε τα υπέρ και κατά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επίλυση διαφορών. Στη Δανία, για παράδειγμα, οι εταιρείε ενίοτε πηγαίνουν από μόνε του στο συνήγορο καταναλωτή και λένε Κάναμε κάτι λάθο. Α προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Στη Φιλανδία υπάρχει τώρα ένα νέο συνήγορο καταναλωτών πριν από δύο εβδομάδε ε, ανέλαβε καθήκοντα. Του μιλήσαμε και ήδη έχουν προκύψει δύο-τρεις υποθέσεις που όπως είπατε χρησιμοποίησε το ενδεχόμενο αυτής της ε, μαζικής ε, ε, αγωγής, συλλογικής αγωγής. Αυτό δημιουργεί νευρικότητα και επομένως κάνει τον παραβάτη να θέλει να προχωρήσει σε διακανονισμό. Σε άλλες χώρες λείπει. Στο Βέλγιο το είχαμε το ίδιο πράγμα. Για τις ενός καταναλωτών, αλλά είναι μία. και είναι η μόνη που μπορεί να κάνει ε, συλλογικέ προσφυγές. Υπάρχει και μια άλλη ε, οργάνωση. Personally think... Ενελικτική επίλυση διαφορών. Άλλη δυνατότητα. Και αν μιλάμε για αυτό το μέσο, συλλογική ένδειξη προστασία χάθηκε μια ευκαιρία με την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Γιατί μιλάμε σε πολλέ περιπτώσει για διασυνορικέ υποθέσει. δεν σταματάνε στα σύνορα, άρα χρειάζεται ένα κατάλληλο πλαίσιο στον κανονισμό Βρυξέλλες 1 που θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα, αλλιώς θα υπάρχει forum shopping και θα υπάρχουν διάφορες. Κοινές θέματα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Uh, κύριε Ολιβέρα, θέλετε και εσείς το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να απαντήσω στα τρία ερωτήματα της κυρίας Ρέντα. Για το μέσο, το εργαλείο. Έχουμε αμφιβολίες που έχουν να κάνουν με διαδικαστικά ζητήματα περισσότερο. Τι θα γίνει, πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα κράτη-μέλη στο σύστημα και εάν το επιλέξουμε τελικά αυτό το εργαλείο, τι δυνατότητες υπάρχουν από πλευράς νομικής βάσης. Γιατί ζητούμε εδώ κάποιες σοβαρές ασφαλιστικές δικλίδες, εχέγγυα, που δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. αυτό μας ανησυχεί τα μάλα. Έπειτα θα θέλαμε να περιοριστεί μόνο στο δικαίωμα καταναλωτών, διότι αλλιώς ε, θα έχουμε ένα ε, μια πολύ ευρύτερη συζήτηση γιατί θα πρέπει να καλύψουμε το σύνολο του ενοχικού δικαίου. We don't have yet an abuse. Και για την ε, κατάχρηση ε, αυτών των διαδικασιών Κάποιες περιπτώσεις είναι ιονή η καταχρήση. Να σας αναφέρω τρεις περιπτώσεις. Στη Γαλλία είχαμε μια υπόθεση για τις κοινωνικές μισθώσεις, κοινωνικές κατοικίες, η εταιρεία ε, προσέφυγε σε σχέση με μια καταχρηστική ρίστα, ρήτρα και είχαν ε, φουσκώσει ε, τους, τα θύματα των εισαγωγικών σε μισό εκατομμύριο. Ενώ ο δικαστής βρήκε τέσσερις μόνο τελικά που επλήγησαν από την εν λόγω ρήτρα. Αυτό είναι ένα κίνδυνο λοιπόν να ε, των ε, διαδίκων. Στην Ολλανδία είχαμε την υπόθεση Λότο, την πολύ διάσημη αυτή υπόθεση, όπου ο διευθυντής του φορέα που συγκέντρωνε τις καταγγελίες από τα 8 εκατομμύρια που, που εισέπραξε, τα μισά τα πήγε σε μια εξωχώρια εταιρεία. Και κάποια από αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει πολύ ακριβά αυτοκίνητα, γιατί είχε ακριβά γούστα. Άλλη μια δεύτερη περίπτωση. Και κάτι που δεν είναι ακριβώς ε, κατάχρηση, αλλά σας δείχνει πώς μπορεί η χρηματοδότηση ε, τρίτο να ε, ωφελήσει κάποιους, ε, όπως ήταν η περίπτωση Mastercard. 40 εκατομμύρια ευρώ ήταν η επένδυση, θα έπρεπε στο τέλος να είχαν πάρει 135 εκατομμύρια. Ως αποζημίωση, όμως, επειδή δεν, δεν είχαν διανεμηθεί πολλά από αυτά τα χρήματα, μπόρεσαν να τα κρατήσουν και έφτασαν στο ένα δις. Δεν ακριβώς κατάχρηση αυτό όπως είπα, αλλά τέλος πάντων βλέπετε τι είδου προβλήματα να με αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, εμπιστατωμένες απαντήσεις. Μια ερώτηση όμως είχα που δεν απαντήθηκε προς την Κομισιόν συγκεκριμένα. Ποιο είναι το επίπεδο αναρμόνιση, Για παράδειγμα, αυτό ο δανό συνήγορο του καταναλωτή στις συστάσει και στην έκθεση συνέχεια, η Κομισιόν προτείνει ε, το opt μοντέλο πιο πολύ. Άρα θα την κρατήσει την πυρηνική βόμβα ως επιλογή ο δανός συνήγορος αν μείνει ε, έτσι η πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Η Κομισιόν, ναι, όπως σας είπα, Μία από τις παραμέτρους ε, που λαμβάνουμε δε όντως υπόψη είναι οι διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Επομένως, όποιο και αν ε, είναι το εργαλείο που θα σχεδιάσουμε στο τέλος, αυτό θα πρέπει να είναι παρκώς ευέλικτο, ώστε να προσφέρει τα απαραίτητα χέγγια αλλά παράλληλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν τους μηχανισμούς ε, συλλογικής ένδικης προστασίας που έχουν ήδη και που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα προσπαθούμε να τον πετύχουμε. Θα προσπαθήσουμε να τον πετύχουμε. Ευχαριστώ. Uh, has the questions of mm, the members been responded to? Ε, υπάρχει κάτι ε, άλλο το οποίο πρέπει να λεχθεί από κάποιους κύριους Διντιέ το ερώτημά μου αφορά την Επιτροπή, γιατί γνωρίζουμε ότι οι διαφορές υπερβαίνουν τα σύνορα και δεν θα πρέπει κράτη-μέλη να ε, σταματήσουν την συλλογική ένδικη προστασία. Δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδι δηλαδή σε αυτούς τους ε, μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας. Δεν ξέρω λοιπόν ε, κατά πόσο οι δικαιοδοσίες σε άλλα κράτη-μέλη μπορούν να δράσουν ή να μην δράσουν. Γιατί οι οικονομικές δραστηριότητες ε, ξεπερνούν τα σύνορα, καθώς και οι διαφορές. Εντάχει από την Επιτροπή, μάλλον ο καθηγητής Βέτ. Επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο στο Βέλγιο εξέδωσε απόφαση γιατί σύμφωνα με, το βελγικό δίκαιο μία ένωση καταναλωτών μπορεί να προβάλλει ένα μηχανισμό συλλογικής προστασίας. Αυτό το αμφισβήτησε το Συνταγματικό Δικαστήριο και είπε ότι αποτελεί παραβίαση της οδηγίας περί Ανέφερε λοιπόν ότι οι ενώσεις καταναλωτών στις χώρες τους μπορούν να προβάλλουν αξιώσει στο Βελγικό Δικαστήριο. Αυτό αναφέρθηκε λοιπόν στην απόφαση του Βελγικού Συνταγματικού Δικαστηρίου όταν αναφέρθηκε στην Οδηγία Υπηρεσιών. Το κατά πόσο ισχύει είναι συζητήσιμο. Επιτροπή. Μικρόφωνο παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή δεν προβλέπει αλλαγές στη, στα μέσα και τους μηχανισμούς του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπως ισχύουν στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν στις συλλογικές αγωγές και προσδίδουν ασφάλεια δικαίου και υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων. Γνωρίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο διευκόλυνσης στις συλλογικές αγωγές διασυνοριακά, σε διασυνοριακές διαφορές δηλαδή. Αλλά ίσως οι συνάδελφοι που εργάζονται επ' αυτού μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ όπως είπα. Ε, βρισκόμαστε σε πρωταρχικό στάδιο, αλλά ε, ασχολούμαστε με την τρέχουσα οδηγία περιασφαλιστικών μέτρων έτσι ώστε οι φορείς που ε, ορίζονται από τα κράτη-μέλη θεωρούνται οι κατάλληλοι φορείς για να προβάλλουν ε, αξιώσεις ασφαλιστικών μέτρων σε άλλα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με διασυνοριακές διαφορές που γίνονται όλο ένα και περισσότερες. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας, ε, ε, ε, έλαβα μια ερώτηση από το κοινό, από τον κύριο Ντάλι σε σχέση με μία έρευνα που διενεργήθηκε σε δεκα κράτη-μέλη σε σχέση με τους ε, μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διενεργήθηκε από ένα επιμελητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να μου πείτε λεπτομέρειες. Ε, εγώ εκπροσωπώ το επιμελητήριο των ΙΠΑ και όπως είπα, οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν οριστεί στη σύσταση της Επιτροπής ακολουθούνται από την οδηγία Injunctions Plus. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η Επιτροπή θα συνεχίσει να ακολουθήσει τη δική της σύσταση έτσι ώστε οι ίδιες δικλίδες ασφαλείας να ισχύουν παντού. Και μετά δηλαδή από την εφαρμογή της οδηγίας ασφαλιστικών μέτρων. Νομίζω μονολεκτική μπορεί να είναι η απάντηση. Θα άρχιζα με το ναι, αλλά ναι ότι θα απαντήσω στην ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Η σύσταση παραμένει και οι αρχές της σύστασης ισχύουν και γι' αυτό ζητούμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές και να τις ενσωματώσουν στα ε, νομικά τους συστήματα. Ίσως ο συνάδελφος μπορεί να πει κάτι περισσότερο για αυτούς τους μηχανισμούς για το μέλλον. Και πάλι μία λέξη. Οι αρχές ισχύουν και ελπίζουμε να τηρηθούν από τους πάντες και την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ως προς το συγκεκριμένο ένδικο μέσο, Ίσως δεν χρειάζεται κάθε φορά να επαναλαμβάνονται οι αρχές. Το ζήτημα είναι πώς θα οριστεί αυτό το μέσον. Γιατί εμείς ε, δεν συντάσσουμε τους, ε, τον κώδικα ε, της αστικής δικονομίας. Απλώς ασχολούμαστε με επιμέρους σημεία δεν χρειάζεται να, αναφέρετε να αναφέρονται αυτά τα μέσα κάθε φορά. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρόντες σήμερα και για τα μέλη να πω ότι θα συναντηθούμε το απόγευμα.